interinstitutional agreement we will have to put also this condition. Θα πρέπει Αγαπητοί συνάδελφοι, να αρχίσουμε. Είναι 3 και 12, αλλά επειδή ο Υπουργό είναι εδώ, θα ήθελα να αρχίσει η συνεδρίαση. Όπως ξέρετε, θα συζητήσουμε με τον Υπουργό Οικονομίας, κύριε Ριμάντα Σάντζος, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, και να του δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει το, πρόβλημα, το πρόγραμμα της λιθανικής Προεδρίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια πολύ καλή παράδοση στα θεσμικά όργανα, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο. Όταν αρχίζει η Προεδρία, Αρχίζουμε τις ε, παρουσιάσεις στη γλώσσα της χώρας. Γι' αυτό σας παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας. Θα μιλήσω λιθανικά. Κυρία Πρόεδρε, ε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή η συμμετοχή μου σήμερα στην συνεδρίασή σας όπως και στις άλλες συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου για να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Λιθανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στην Επιτροπή σας οι προτεραιότητες έχουν να κάνουν με την πολιτική συνοχή και την μακροπεριφερειακή στρατηγική. Ως Λιθουανός Υπουργός Οικονομίας είμαι υπεύθυνο ε, για την πολιτική σε αυτούς τους τομείς η κατάσταση φυσικά δεν είναι η ίδια σε όλες τις χώρες αλλά θεωρώ ότι αυτό αυξάνει τη σημασία των θεμάτων που σχετίζονται με την περιφερειακή πολιτική τα οποία θα γίνουν ακόμη πιο σημαντικά κατά τη διάρκεια της Λιφανικής Προεδρίας. Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ με σας τις ε, απόψεις μου για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα κοινά θέματα της επόμενες, τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Είναι πρώτη φορά που η Λιθουανία ε, προεδρεύει του Συμβουλίου. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ούτως ώστε η Προεδρία να διεξαχθεί υπό το ελάχιστο κόστος, αλλά να είναι επίσης ε, αποτελεσματική και να επιδιώξει να επιτύχει αποτελέσματα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα. Οι τρεις προτεραιότητες της Προεδρίας μας είναι αξιοπιστία, ανάπτυξη και διαφάνεια στην Ευρώπη. Οι καλύπτουν ε, όλα τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την Ένωση. Είμαι ε, πεισμένο γι' αυτό. Σε κάθε τομέα, κάθε υπουργό έχει βεβαίως ε, τις δικές του προτεραιότητες. ω υπουργό οικονομία και Προεδρεύων του ΕΚΟΦΗΝ, πρώτα απ' όλα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει αξιοπιστία της Ευρώπης ε, έναντι των χρηματαγορών. Η ανάπτυξη της Ευρώπης επίσης είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα για όλους τους πολίτες, σε όλους τους τομείς πολιτικής. Και επίσης ε, θέλουμε η Ευρώπη να είναι διαφανής. Χθες ε, προέδρεψα του πρώτου Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ και με χαρά καλωσόρισα δύο χώρες την Κροατία που έγινε το 28ο μέλος της Ένωσής μας και την Λετωνία. Ε, καλωσορίσαμε την Λετωνία ε, στη ζώνη ευρώ και γι' αυτό χρειάστηκε να εγκριθεί τα κατάλληλα νομοθετήματα για να μπορέσει να νομοθετήματα για να μπορέσει να ε, ενταχθεί η Λετωνία ε, και για να μπορέσει να ξεκινήσει το λαμπρό μέλλον της ε, στην Ευρωζώνη. Η Ένωση γενικά έχει ένα τεράστιο εσωτερικό δυναμικό που δεν έχει αξιοποιηθεί. Αυτό πρέπει να το αποδείξουμε ε, σε όλες τις περιοχές του κόσμου που μας περιβάλλουν. Η Προεδρία μας ε, διεξάγεται σε μια περίοδο ε, όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις. Η δημοσιονομική εξυγίανση είναι αναγκαία για να επανέλθει η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών οικονομίες της χώρας μας. Πρέπει να αναθεωρηθούν για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και για να αυξηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στον κόσμο. Αλλά κύριος στόχος μας είναι η ανάπτυξη των οικονομιών μας, η οικονομική αύξηση η ημερήσια διαταξή μας καλύπτει τις χρηματαγορές, ε, την ε, φορολογία, άλλους τομείς και την ε, νομοθεσία που χρειάζεται. Για να επιτύχουμε την ανάπτυξη χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέσα. Η πολιτική της συνοχής είναι ένα από τα κύρια όργανα προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα να αναφερθώ στις συγκεκριμένες προτεραιότητές μας στον τομέα της πολιτικής συνοχής. να συζητήσουμε τώρα τις περαιτέρω προτεραιότητες σε λεπτομέρεια της Προεδρίας μας στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχής είναι στη καρδιά της ε, προσπάθειας ανάπτυξης και απασχόλησης. Όχι μόνο συμβάλλει στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων που ακόμη έχουμε, αλλά έχει επίσης επίδραση συνολικά στην οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο των διαφόρων περιφερειών όπου δεν υπάρχει ήδη επαρκές ε, δυναμικό ανάπτυξη αλλά συνολικά για την Ευρώπη. Η ενιαία αγορά είναι η βάση της Ένωσης. Ένας από τους λόγους γιατί η πολιτική συνοχή είναι αναγκαία, ένας λόγος γιατί χρειαζόμαστε επίσης ε, περιφερειακή πολιτική, είναι να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς για να διασφαλιστεί πρέπει να ξέρουμε πού και πότε να παραχθούν αγαθά και υπηρεσίες και πού και πώς να διατεθούν. Πρέπει και η προσφορά και η ζήτηση να λειτουργούν σωστά. Η προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής είναι επίσης προφανής και έχει αυξηθεί στους ε, τόσο δύσκολους καιρούς που περνάμε. Για μερικές χώρες ήταν το κύριο όργανο για να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση, η οικονομική, η χρηματοπιστωτική κρίση. Η χώρα μου, η Λιθουανία, δεν αποτελεί εξαίρεση. Τα διαθροτικά ταμεία μας βοήθησαν ιδιαίτερως για να καλύψουμε την καθυστέρησή μας όταν δεν υπήρχε δυνατότητα δημόσιας εθνικής χρηματοδότησης. Και εξακολουθεί να μας βοηθάει για να ξεπεράσουμε ε, την δυσχερή κατάσταση στην οποία ήμασταν. Και υπάρχουν και άλλες χώρες σε αυτήν την κατάσταση. Πολλές. Ιδιαίτερα μεταξύ των χωρών που εντάχθηκαν από το 2004 και εντεύθαν. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, να ενισχύσουμε τις εξαγωγές, τις επενδύσεις, να βελτιώσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα και τέλος να μειώσουμε την ανεργία. Αυτοί είναι οι στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν με την ε, πολιτική συνοχής. Γι' αυτό δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μεγάλες καθυστερήσεις στην εφαρμογή συγκεκριμένης δράσης. Δηλαδή πρέπει να εγκριθούν τα νομοθετήματα που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Λαμβάνοντα υπόψη ότι, ότι την 1η του 14 θα ε, τεθούν σε ισχύ οι νέε ε, πολιετής δημοσιονομικέ προοπτικέ. Αυτή είναι η κοινή μα πρόκληση λοιπόν, χωρίς καθυστερήσει, χωρίς πισωγυρίσματα, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, ούτω ώστε τα εργαλεία τη πολιτική συνοχή να μπορέσουν να αρχίσουν να λειτουργούν. Πρέπει να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις για να αρχίσει να ισχύει μετά την έγκρισή του ο νέος κανονισμός για την πολιτική συνοχή. Αυτό, αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα σε αυτό το τομέα. Θα πρότεινα εδώ, επειδή ακριβώς ε, ο χρόνος επήγει, να μην ασχοληθούμε με λεπτομέρειες. Να επιδιώξουμε την επίτευξη του κοινού στόχου που είναι σαφέστατος, γιατί είναι σαφέστατο ότι πρέπει να απελευθερώσουμε πάνω από 300 δις ε, διαφορετικής βοήθειας για τις επιχειρήσεις, για τους ανέργους, για αυτούς που επιδιώκουν να βελτιώσουν ε, την εκπαίδευσή τους, για τη βελτίωση των υποδομών, όπου δεν επαρκούν. Οπότε, πρέπει επίσης να τονίσω ότι ε, χρειαζόμαστε και την δευτερογενή νομοθεσία που δεν μπορεί να ε, συζητηθεί πριν καταλήξουμε όσον αφορά τον βασικό κανονισμό. Άρα ο χρόνος πιέζει ιδιαίτερα. Ένα άλλο θέμα είναι λοιπόν αυτός ο γενικός κανονισμός. Είναι φυσικά από τα θέματα που μας απασχολούν. Πιέζει ο χρόνος Πρέπει να απαλύνουμε τις επιπτώσεις της κρίσης για αρκετές χώρες που χρειάζονται την βοήθειά μας περισσότερο από άλλες. Έχουμε λοιπόν ε, τη βούληση για να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των συνομοθετών για το θέμα αυτό το ταχύτερο. Διότι είναι πράγματι επίγον, πραγματικά επίγον. Στη νέα περίοδο, περίοδο προγραμματισμού θα επιδιώξουμε να αναπτύξουμε την μακροπεριφερειακή στρατηγική της Ένωσης, ιδιαίτερα για την περιοχή της Βαλτικής. Η πρώτη μακροπεριφερειακή στρατηγική της Ένωσης ε, προτάθηκε και εξακολουθεί να επιτηρείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με βάση τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Προεδρία θα οργανώσει συζητήσεις στο Συμβούλιο για να αναθεωρηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε όλες τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές που έχουμε ενώπιόν μας. Και κυρίως θα μας απασχολήσει το θέμα της προστιθέμενης αξίας που μας παρέχει αυτή η στρατηγική. Γιατί ορισμένες φορές δεν διαπιστώνουμε τέτοια προστιθεμένη αξία στις μακροπεριφερειακές μας στρατιστικές, στρατηγικές. Και αναγνωρίζω ότι στον τομέα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντική κινητήριος δύναμη. Προσβλέπουμε λοιπόν στη γνώμη, στη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η κοινοβουλευτική διάσταση με τη συμμετοχή και των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι πολύ σημαντική. Και με χαρά ανακοινώνω ότι στις 11 και 12 Νοεμβρίου στο Βίλνιους θα λάβει χώρα το 4ο ετήσιο φόρουμ για την ε, ενωσιακή στρατηγική στην περιοχή της Βαλτικής. Να συζητήσουμε λοιπόν τα κοινά προβλήματα και ε, με χαρά σας προσκαλούμε κυρία Πρόεδρε εσάς και όσους συναδέλφους σας θέλουν να συμμετάσχουν για να συζητήσουμε αυτό το θέμα της προστιθέμενης αξίας που είναι απαραίτητο στοιχείο κάθε στρατηγικής, άρα και αυτής. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός, μια άλλη σημαντική εκδήλωση που θα γίνει επίσης τον Νοέμβριο θα είναι η άτυπη συνάντηση των Υπουργών που είναι υπεύθυνοι για την πολιτική συνοχή. Θα λάβει η χώρα στις 26 Νοεμβρίου. Θα είναι μια δυνατότητα να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα της προετοιμασίας για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Αυτή η άτυπη υπουργική συνάντηση θα ήταν το κατάλληλο βήμα για να κάνουμε πολύ χρήσιμες συζητήσεις με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό και πάλι σας προσκαλώ θερμά να συμμετάσχετε σε αυτήν τη σημαντική συνάντηση. Επίσης, τελευταίο σημείο, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε την εργασία και τα επιτεύγματα των προηγούμενων προεδριών. Θέλουμε να υπάρχει μια συνέχεια στην εργασία των προεδριών και εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την εργασία της Ιρλανδικής αλλά και των προηγουμένων προεδριών που προετοίμασαν αυτή τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Επίσης, Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως στην ε, Επιτροπή σας. Τους εισηγητές, αλλά και η δική σας ε, προσωπική συμβολή, κυρία Πρόεδρε, ήταν πολύ σημαντική. Σας διαβεβαιώ ότι η αποτελεσματική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι συνομοθέτης, θα είναι η προσωπική μου προτεραιότητα. Όχι μόνο βέβαια με την Επιτροπή σας, αλλά και με άλλες. Και αναλαμβάνω λοιπόν την προσωπική ευθύνη να διασφαλίσω ότι θα διεξαχθεί ομαλά αυτή η συνεργασία γιατί και εγώ και οι συνεργάτες μου καταλαβαίνουμε την αυξανόμενη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, αντανακλά την ε, συνολικότερη αύξηση σημασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι του χρόνου θα έχουμε ευρωεκλογέ και ελπίζω η προεκλογική εκστρατεία να μην είναι εμπόδιο αλλά ένα επιπλέον κίνητρο για να γίνουν πολύ παραγωγικές εργασίες και συζητήσεις μεταξύ μας. Η ομάδα μου, οι συνεργάτες μου έχουν ήδη αναλάβει τις διαπραγματεύσεις από τους Ιρλανδούς συναδέλφους. Έχουν ήδη ξεκινήσει τριμερίς τριμερείς διάλογοι. Ήδη τώρα τον Ιούλιο θα έχουμε άλλη μια σειρά τριμερών διαλόγων για την περιφερειακή πολιτική από αύριο, ήδη αύριο. Ήδη προγραμματίζουμε μια ιδιαίτερα απαιτητική ημερήσια διάταξη για τον Σεπτέμβριο. Αν υπάρχουν τεχνικά θέματα, μπορούμε βεβαίως να διοργανώσουμε συζητήσεις ήδη τον Αύγουστο σε τεχνικό επίπεδο. Είμαστε προπαρασκευασμένοι, είμαστε διατεθειμένοι να προωθήσουμε τα θέματα αυτά. Προσβλέπω λοιπόν στη συνέχιση της κοινή μας προσπάθειας για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες μας και τους λαούς μας. Σας ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτήν τη δυνατότητα που μου δώσατε να μοιραστώ τις απόψεις μου μαζί σας. Με πολύ χαρά θα ακούσω τις δικές σας απόψεις για θέματα περιφερειακής πολιτικής, γιατί φυσικά η Προεδρία παίζει ένα ρόλο ε, επιδιαιτητή στις συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο. Θα επιχειρήσουμε να είμαστε έντιμοι διαμεσολαβητές να οικοδομούμε συμβιβασμού. Για να γίνει όμω αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα δίκτυο σχέσεων, καλή συνεργασία με όλου του εμπλεκομένου και του υπουργού και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση με του υπουργού ε, οικονομία και με τι κυβερνήσει, άρα θα θεωρούσα των κρατών μελών αλλά επίση και με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των, επιτροπών δηλαδή με τι οποίε ασχολούμαι. Προσβλέπω λοιπόν σε αυτή την καλή συνεργασία. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας, τις θέσεις σας, για να βελτιώσουμε ουσιοδός τη συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Θα λέγω ότι είναι ενθαρρυντικά αυτά που μας λέτε. Ελπίζω κι εγώ ότι θα έχουμε μια καλή Προεδρία και ότι θα αλληλοβοηθηθούμε στο τελικό μας στόχο που είναι να προχωρήσουν οι πολιτικές μας όπως είπατε για η Ευρώπη τη χρειάζεται την ανάπτυξη. Τώρα συζήτηση. Οι συντονιστές πρώτα. Εκ μέρους του ΕΛΚ ο Λαμπέρ Φανίστερόι. Ευχαριστώ. Ναι, πολύ σύντομα εκ μέρους του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που ήρθατε. Σας ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων. Φυσικά, οι προσδοκίες μου είναι μεγάλες από την Προεδρία σας, από τη συνεργασία μαζί σας. Σήμερα το πρωί ψηφίσαμε διάφορα θέματα που είχαν προχωρήσει από την προηγούμενη Προεδρία και πολλές φορές και το Συμβούλιο και η Επιτροπή τα στήριξαν. Η προσέγγιση είναι θετική και τη χρειαζόμαστε αυτή τη θετική προσέγγιση γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε αν μη τι άλλο όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι μέσα στο πακέτο, στο ίδιο πακέτο δηλαδή, και ως συνομοθέτες πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Υπάρχουν δυσκολίες, το αναφέρατε και εσείς, το θέμα της ρεσιμότητας, το θέμα των επιδόσεων, το θέμα της προχρηματοδότησης, του ποσοστού κλπ. Ένα σημείο θα θίξω. Είπατε, 26 Νοεμβρίου θα υπάρξει μια άτυπη διάσκεψη υπουργών. Αν λοιπόν με ρωτήσετε τι περιμένω εγώ από αυτήν, θα έλεγα έρευνα και ανάπτυξη, ο συνδυασμός αυτός. Έχουμε το πρόγραμμα ορίζοντας 2020 με 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναθερούμε την πολιτική συνοχής Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις με τις οποίες έχουμε συμφωνήσει, το στρατηγικό πλαίσιο, συνεργασία κλπ. Διάφορα εργαλεία δηλαδή, με τα οποία με τη θεματική συγκέντρωση μπορούμε να δώσουμε τεράστια όθηση στις περιφέρειες και στις χώρες μέλη εκείνες που επιλέξουν να συνδυάσουν την χρήση των ικανοτήτων των ανθρώπων και να συμπεριλάβουν τον ιδιωτικό τομέα της επιχειρήσης. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί το δημόσιο, εντάξει, μπορεί να είναι σημαντικό, αλλά σήμερα δεν έχουν χρήματα για θέσεις απασχόλησης. Στις περισσότερες χώρες πάει, έχουν εξανεμιστεί. Οπότε αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να μην καθόμαστε και μιλάμε μεταξύ μας. Εντάξει, ευχαριστούμε και για την πρόσκληση, θα έρθουμε αλλά να μην καθόμαστε και μιλάμε μεταξύ μας με αυτούς που είναι ήδη για τη συνοχή, αλλά να υπάρξει μια υπουργική διάσκεψη με εκείνους που κάνουν την έρευνα και την ανάπτυξη, που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, και να τους φέρουμε πιο κοντά στην απασχόληση και την καινοτομία. Δηλαδή βγείτε λίγο από αυτούς τους πυλώνες, γιατί είναι σαν να δουλεύουμε έτσι με, με πυλώνες. Αυτό που έχω ακούσει εδώ στο Κοινοβούλιο είναι να δίνουμε τόσα για έρευνα και τεχνολογία. Όχι. Τα κονδύλια τα έχουμε, αλλά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά και αυτό ακριβώς είναι που προτείνουμε με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Στο κείμενό σας διάβασα ότι υπάρχει αυτή η προσέγγιση η πιο ολοκληρωμένη. Θα καινοτομήσετε ή θα ακολουθήσετε το δρόμο που έχουν ήδη χαράξει οι πιο παλιοί. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε στην κάθε ερώτηση χωριστά, κύριε Υπουργέ, ή συνολικά. Ωραία. Θα ακούσουμε την επόμενη ερώτηση. Η Κωνσταντ Σακρέλ, εκ των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Ντανούτα. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πολύ. Εδώ είμαι. Χαίρομαι πολύ που είναι δυνατόν να έχουμε τόσο ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για την επόμενη Προεδρία Θα έλεγα ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη, διότι η πρώτη διάλογη, η τριμερής διάλογη η προεδρία ήταν ε, ευχάριστα δυναμική και ήδη έχουν σημειωθεί κάποιες πρόοδοι. Επιτρέψτε μου να είμαι ειλικρινής, είναι τώρα η τέταρτη προεδρία με την οποία συνεργάζομαι ως εισηγήτρια για το Γενικό Κανονισμό και δεν ήσαν όλες οι προεδρίες τόσο ευέλικτες, τόσο ανοιχτές στους τριμερείς διαλόγους. Θεωρώ ότι είναι θετικό επίσης το ότι είναι πρώτη φορά που διαπραγματεύουμε με μια μεικτή ομάδα. Δηλαδή μια ομάδα όπου από πλευράς προεδρίας υπάρχουν πολύ περισσότερες γυναίκες ειδικοί από τις προηγούμενες προεδρίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί να καταδεικνύει ότι τόσο πιο μικτές ομάδες είναι πραγματικά καλύτερες. Μα ναι, και εμείς είμαστε βέβαιως ε, μεικτή ομάδα, ο Λάμπερτ και εγώ. Ήδη από τη Δανέζικη Προεδρία έχουμε πει ως Κοινοβούλιο επανειλημμένα και θα το ξαναπούμε το Σεπτέμβριο είναι ότι σε όλες τις διαπραγματεύσεις που έχουν κάνει οι προεδρίες με το Κοινοβούλιο για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, 80% των διαπραγματεύσεων είχαν να κάνουν άμεσα με την πολιτική συνοχής και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να είναι η διαδικασία του πολιετούς πλαισίου αλλά θα έπρεπε να ήταν ε, στο πλαίσιο της συναπόφασης δηλαδή να αντιμετωπίζονται ισότιμα τα δύο θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Και αυτό που μας ε, απομένει τώρα, το περίπου 5% που δεν μπορέσαμε να το βάλουμε στον γενικό κανονισμό, είναι όπως είπε και ο Λάμπερτ, είναι τα πράγματα, η μακροαιρεσιμότητα, το αποθεματικό, η, η προχρηματοδότηση, η συγχρηματοδότηση. Και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τον Φεβρουάριο νόμιζαν ότι είχαν αποφασίσει. Αλλά είναι θέμα συναπόφασης. Ίσως λοιπόν να μην το επιθυμούσαν οι δικοί σας όταν ανέλαβαν την Προεδρία να χρειαστεί να πιέσουν τους υπόλοιπου αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων για να επιτευχθούν συμβιβασμοί. Ελπίζω όμω να το κάνουν και να επιτευχθούν συμβιβασμοί. Είναι βεβαίω πρόκληση για ένα κράτο μέλο που πρώτη φορά αναλαμβάνει την Προεδρία και που δεν είναι βέβαια από τα μεγαλύτερα κράτη της Ένωσης είναι σίγουρα μια ιδιαίτερη πρόκληση να βοηθήσετε να επιτευχθεί λύση. Πιστεύω όμως ότι τα 500 εκατομμύρια πολίτες της Ένωσής μας θα ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι αν το επιτυγχάναμε. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει μεγάλη σημασία να καταλήξουμε το Σεπτέμβριο σε συμβιβασμούς. Γιατί αυτό το μέσο είναι νέο και μοναδικό μέσο επενδύσεων, είναι το μοναδικό που έχει αυτή τη φορά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό την 1η πρώτου 14 να είναι έτοιμο. Εάν το επιτύχουμε και για την προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογέ που είναι λίγο μετά και βεβαίω για την επανεκλογή τη Κομισιόν είναι ένα πολύ καλό μήνυμα ότι θα έχουμε επιτύχει να προωθήσουμε αυτή την πολιτική. Δεν είναι ερώτημα αυτό που σας θέτω, είναι επιθυμία να το επιτύχουμε από κοινού και ελπίζω να συνοηθούμε και να καταλήξουμε σε σκόπιμο αποτελέσμα το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εκ το μέρους των φιλελευθέρων υπάρχει κάποιος που θέλει κάτι να πει. ECR μήπως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ εδώ. Και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις τώρα στην αρχή της Προεδρίας που μπορούμε να αλληλοενημερωθούμε. ενημερωθούμε. Εγώ είμαι από την Τσεχία, πρέπει να ξέρετε. Που σημαίνει ότι έχω ήδη περάσει από την Προεδρία και είναι, πιστεύω, μεγάλη τύχη για κάποιον να μπορεί να συνεισφέρει στο μέλλον της Ευρώπης. Συμφωνώ με την Κωνσταντς. Και η δικιά μου πολιτική ομάδα στηρίζει την ιδέα των μεικτών ομάδων. Η ατμόσφαιρα είναι πάντα πιο ευχάριστη, η συνεργασία πηγαίνει καλύτερα κλπ. κλπ. Όσον αφορά τώρα τις χώρες που αργότερα εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο συμβιβασμός αυτός που θα συμφωνηθεί το φθινόπωρο είναι πολύ σημαντικός. Είμαστε λίγο πριν τις επόμενες ευρωεκλογέ και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα βγούμε και θα στηρίξουμε τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες μπροστά στο εκλογικό μας σώμα αν δεν έχουμε να τους προσφέρουμε και κάτι ενδιαφέρον στις προτεραιότητές μας. Οπότε, Ευχαρίστως να αποτελέσω το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε εσά και τους αξιωματούχους της χώρας μου, με τους οποίους θα μπορέσετε να έχετε επαφές. Κάτι πολύ σημαντικό για μένα είναι το αποτέλεσμα που πέτυχα στην προηγούμενη δουλειά μου, που ήμουν δήμαρχος δηλαδή. Οπότε, για μένα και για τους συναδέρφους μου πρέπει να ξέρετε ότι το μέλλον της Ευρώπης και ο τρόπος που θα εξελιχθεί η οικονομία μας εξαρτάται κατά πολύ από το πόσο ελκυστικές είναι οι πόλεις μας, οι μεγάλες πόλεις της χώρας μας. <clears throat> Ελπίζω και εσείς να λάβετε υπόψη σας αυτό το στοιχείο και να είναι και για σας προτεραιότητα μια τέτοια πολιτική υπέρ των πόλεων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Και εμεί ευχόμαστε να πάει όσο γίνεται καλύτερα η Προεδρία σας. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που βέβαια είναι πολύ σημαντική ακριβώς επειδή βρίσκεστε στο τέλος της πολιτικής που έχει ήδη αρχίσει την προηγούμενη χρονιά μέσα από διαδοχικές προεδρίες και πια σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που θα διασφαλίσει τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, που είναι πολύ βασικές πολιτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Ιδιαίτερα, μάλιστα, σε σχέση με τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει βάλει πολλές ελπίδες στην μελλοντική πολιτική συνοχής υπήρξε η ενίσχυση των μέσων εδαφικής συνεργασίας για παράδειγμα και αποφασίσαμε 7% του Ταμείου Συνοχής να πάνε ακριβώς εκεί. Η πρόταση βέβαια της Κομισιόν δεν έφτασε μέχρι εκεί αλλά τουλάχιστον υπήρχε κάποια ενθάρρυνση. Τελικά έγιναν διάφορες διαιτησίες οι οποίες όμως μας απογοήτευσαν το Φεβρουάριο που πέρασε τελικά η πολιτική αυτή εδαφική συνεργασίας, που για το μέλλον θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κατέληξε να πρικοδοτηθεί με ελάχιστα κονδύλια. Κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Και γιατί, γιατί το είπατε κι εσεί υπάρχουν διαδικασίες που προχωράνε, οι χώρες τη Βαλτική είναι πολύ καλό που την πρωτοβουλία αλλά η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να παραμείνει στη Βαλτική, πρέπει να είναι μια διαδικασία από την οποία να υποφεληθούν όλοι οι πολίτες στην Ευρώπη και να υπάρξει έτσι παντού καλύτερη συνεργασία. Εσείς είπατε ότι αυτό το θέμα σας ενδιαφέρει. Σας ενθαρρύνω λοιπόν να συνεχίσετε με την πρωτοβουλία αυτή, ώστε να προετοιμαστεί τον μέλλον των πολιτικών αυτών με έναν ενισχυμένο ρυθμό. Αυτό ίσως σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε όλοι σας την επιρροή στο Συμβούλιο ώστε η δαφική συνεργασία να προχωρήσει, να χρησιμοποιηθεί η ευελιξία που συζητάμε για το μέλλον του προπολογισμού και να βρεθεί και ο τρόπος να εφαρμοστεί η ευελιξία αυτή, τα κονδύλια δηλαδή που χρειάζονται. Να λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία μπορείτε να φροντίσετε κατά τη διάρκεια του, της Προεδρίας σας και εσείς. Ευχαριστώ. Also, καταρχά äh, ich möchte antworten καταρχάς να απαντήσω ότι και εγώ χαίρομαι που έχουμε μεικτή ομάδα είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας, γιατί έχουμε πολλές ειδικού και στο Υπουργείο Οικονομίας, αλλά και σε άλλα Υπουργεία. Οι κυρίες αυτές είναι πολύ μορφωμένες. καταρτισμένες αλλά δυστυχώς ε, τα γερμανικά δεν είναι η πρώτη μας ε, γλώσσα, οπότε μάλλον... Θα περάσω στα αγγλικά για να συνεχίσω και να εκφράσω τις απόψεις μου για, το άκρος, για τα άκρο σημαντικά προβλήματα και τις παρατηρήσεις που κάνατε. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές για τις ερωτήσεις που έθεσαν και τη στήριξή τους για την Προεδρία μας. Είναι πολύ ευχάριστο να ακούω ότι ήδη θεωρείται ότι είμαστε αποτελεσματικοί, παρόλο που πέρασαν μόνο μια-δυο μέρες το μήνα Ιούλιο. Και μόνο εδώ και λίγες μέρες έχουμε αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου. Δεν αληθεύει ότι πάντοτε η Προεδρία αφήνει το σημάδι, του το της και μπορεί να επηρεάσει και τις απόψεις στο Συμβούλιο. Πρέπει βεβαίω να αναζητούμε πάντοτε συμβαστικέ λύσει και διεξόδου. όμως, εγώ και η ομάδα μου σε κάθε περίπτωση, όλοι μου οι συνεργάτε, καταλαβαίνουμε απολύτω τη σημασία των της πολιτικής συνοχής, της εδαφικής συνεργασίας και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βρούμε την καλύτερη πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για το μέλλον. Βεβαίως, όπως προανέφερα, στόχος είναι να φτάσουμε σε συμβαστικές λύσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα. Το πλέον εφικτό για πολλά πράγματα θα είναι ο Σεπτέμβριος. αλλά σε αυτή τη συνεδρίαση μόλις μάθαμε ότι έχετε ήδη ψηφίσει στην Επιτροπή σας για τόσα σημαντικά ζητήματα, με θετικό μάλιστα, μάλιστα αποτέλεσμα και αυτό ήταν ευχάριστη είδηση για μένα και για όλη μου την ομάδα. Ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Νομίζω ότι εδώ μια πραγματική ευκαιρία όλα να προχωρήσουν. Για να μην φτάσουμε στα τέλη Νοεμβρίου τελευταία στιγμή να πιεζόμαστε. Όντι, σε ευχαριστώ για, τις, για τα καλά σου λόγια και την πρόταση να αναλάβεις και εσύ ο συνεργάτης μου στην ομάδα μας μέσω της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Έχουμε σχεδόν τέλειες σχέσεις με όλες τις κυβερνήσεις και των 28 κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του δικού μου βεβαίως στο ΕΚΟΦΗΝ ε, είμαστε σαν οικογένεια. Βεβαίω, οι πολιτική συνοχή δεν είναι απλώ και μόνο αρμοδιότητα των Υπουργών Οικονομικών. Έχουν όμω σημαντικό λόγο στον καθορισμό τη πολιτική αυτή. Να σα πω και ένα μυστικό εδώ. Ότι σε ένα από τα συμβούλια ΕΚΟΦΗΝ προτάθηκε να γίνει συζήτηση για την πολιτική συνοχής και ο Επίτροπος Χάν το πρότεινε αυτό. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η ιδέα και θα δω πώς θα προγραμματιστεί η συζήτηση συγκεκριμένα. Δεν ξέρω ακόμη τις ακριβείς ημερομηνίε και το ακριβές χρονοδιάγραμμα, αλλά είναι καλή ιδέα. Είναι καλή ιδέα και το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ να μελετήσει και αυτό το σκέλος των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τώρα να στραφώ στις ε, πιο σημαντικέ ερωτήσει που άπτονται των αρμοδιοτήτων μου. Ε, Λαμπέρτ, οι δικέ σου ερωτήσει είναι κυρίω, Συμφωνώ απολύτως. Τα εργαλεία της πολιτική συναρχή πρέπει να ανανεωθούν. Χρειάζεται να αναζωογονηθούν και με διαφορετικούς μάλιστα τρόπους, από διαφορετικούς τομείς κάποια πράγματα θα μπορούσαν να συνδυαστούν, ώστε να έχουμε αποτέλεσμα από σχέσεις συνεργασίας. Θα μπορούσαμε να μετατοπιστούμε από το σύστημα δωρεών ή επιδοτήσεων σε οικονομικά, δημοσιονομικά εργαλεία. Αυτό μας αφήνει με καλές πρόπτικες για το μέλλον. Στη χώρα μου, επί παραδείγματι, και ξέρω ότι και στην ευρύτερη περιοχή της Βαλτικής, διότι οι υπουργοί των χωρών της Βαλτικής συναντώνται συστηματικά, όλο ένα και συχνότερα από ότι με τις υπόλοιπες χώρες, για την ευρύτερη γεωγραφική ζώνη της Βαλτικής. Συζητούμε τα θέματα αυτά λοιπόν, σε επίπεδο υπουργών, και είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να υπάρξει μια ε, σημαντική μετατόπιση στο επόμενο διάστημα δημοσιονομικών προοπτικών από τις απλές επιδοτήσεις που δεν θα είναι ποτέ ιδιαίτερα αποτελεσματικές στις επιδοτήσεις συν, δηλαδή το συνδυασμό και με άλλους πόρους. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα γνωρίζετε την πρόσφατη μελέτη που εκπώνησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και συζητήθηκε σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, αλλά και στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ, σε αυτό το σχηματισμό του Συμβουλίου. Μόλις χθε το συζητήσαμε υπό τη δική μου Προεδρία και αποφασίσαμε ότι η Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΕΚΟΦΗΝ θα ασχοληθεί με την βέλτιστη δυνατή υλοποίηση των νέων ιδεών. Όλοι όμως ήδη έχουν κατά νου ότι ο συνδυασμός των διαφορετικών ταμείων και κονδυλίων, των συστημάτων τους, μαζί με δημόσια κονδύλια, πανευρωπαϊκά, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και από άλλες τράπεζες ανάπτυξης που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, μαζί με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, βέβαια, που είναι ένας από τους σημαντικότερους ε, ε, συμβάλλοντες και χορηγούς στην ευρύτερη περιοχή της Βαλτικής μαζί με ιδιωτικέ ε, χρηματοδοτήσεις και τις εταιρικέ σχέσεις δημοσίου-ιδιωτικού ε, τομέα που είναι από τα πλέον σημαντικά εργαλεία και το μελετούμε αυτή τη στιγμή προσεκτικά. Καταλαβαίνουμε ήδη ότι οποιοδήποτε σφάλμα διαπράξουμε τώρα μπορεί να είναι αποφασιστική σημασία. Γι' αυτό Προχωρούμε κάπως αργά, αλλά είμαστε προσεκτικοί. Θα δούμε λοιπόν στην επίσημη σύνοδο για την πολιτική συνοχή στο Βίλνιος κατά πόσον αυτό δεν θα αποτελέσει μια από τις πρώτες προτεραιότητες που θα συζητήσουμε. Μιλάμε για το αύριο της πολιτικής συνοχής. Σαφώς πρέπει να αλλάξουμε τη στάση μας. Δεν μπορούμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό να τον αντιμετωπίζουμε σαν ε, μια αγελάδα από την οποία μπορούμε να αρμέγουμε με μονάδες. Αλλά έχουμε εργαλεία στα χέρια μας. Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε τον τροχό. Τα χρήματα, τα κονδύλια που διαθέτουμε πρέπει να τα ε, φροντίσουμε να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε γενικές γραμμές οι πόροι διαρκώς κλείπουν. Ε, σιγά σιγά θα φθήνουν και την ερχόμενη επταετία. Αυτές είναι οι απαντήσεις μου. Και ανυπομονώ για τις επόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε ο κύριος Όλμπριχτ. Ευχαριστώ Υπουργέ. Σας εύχομαι κάθε τύχη στο εξάμεινο της Προεδρίας σας. Είμαι από την Πολωνία και μιλάμε για μια χώρα αρκετά μεγάλη ως προς τις δυνατότητές της και τα κονδύλια που της ε, απευθύνονται. Έχω όμω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Από πολιτική ε, άποψη, τι γίνεται, είπατε να δράσουμε στο δυνατόν συντομότερα. Αλλά πρώτα, σύμφωνα με το ψήφισμά μα, χρειαζόμαστε πολιτική συμφωνία μέσω τη διαδικασία τη συναπόφαση. Έπειτα υπάρχει συμφωνία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Μετά έρχεται η ψηφοφορία για το Γενικό Κανονισμό Πολιτική Συνοχή που προαπαιτεί την γενικότερη συμφωνία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε σήμερα αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι σχέδια έχετε. Πότε θέλετε το κείμενο για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο να αποσταλεί στο κοινοβούλιο, για, να παραπεμφθεί στο κοινοβούλιο για προσέγγιση. Ξέρω ότι είπατε ω το δυνατόν συντομότερα, το άκουσα, αλλά τι ε, συγκεκριμένο πρόγραμμα έχετε, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, διότι όλο αυτό θα καθορίσει τι διαπραγματεύσει ε, τη αναπόφαση. Εάν πρόκειται για κάτι που δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν είναι προγραμματισμένο, ε, τα πάντα θα, θα, θα μετατοπιστούν ανάλογα με αυτό. Η Σύνοδος των Υπουργών τον Νοέμβριο θα είναι πριν την ψηφοφορία ή μετά. Εάν είναι πριν θα αλλάξει το αντικείμενο, αν είναι μετά θα αφορά την υλοποίηση. Έπειτα, για να είμαι βέβαιος ότι σας κατάλαβα, αναφέρατε στην ομιλία σας ότι βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο 2007-2013. Δεν συζητάμε όμως μόνο το 2014-2020, συζητάμε και το 2007-2013. Ας ε, σκεφτούμε την έκθεση του κ. Βλάσσακ, που νομίζω ότι έφυγε Πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν είναι όμως το τελευταίο τέτοιο ζήτημα που εξετάζουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Και πριν το τέλος του 2013 θα μπορεί να ληφθεί μια δύσκολη, μια σκληρή απόφαση. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για αυτά που επίκυνται. Τι να αναμένουμε στην Επιτροπή μας. Διότι τώρα έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ, υπερβολικά ίσω το 2014-2020. Αλλά πρέπει να τοποθετηθούμε και για άλλα ζητήματα που αφορούν την πολιτική συνοχή με κάπω διαφορετικές διαδικασίες, διότι το 2013 ήταν διαφορετικό, η συναπόφαση ήταν διαφορετική. Εμείς θέλουμε να σας διευκολύνουμε, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε αμέσω τι να περιμένουμε από την Προεδρία σα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε τον Υπουργό που είναι εδώ. Και εγώ ως Ιρλανδός βουλευτής θέλω να τον ευχαριστήσω για τα ευγενικά του λόγια για την Προεδρία μας που μόλις τελείωσε. Νομίζω ότι μπορούμε ως Ευρωπαίοι να χαιρόμαστε για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Το γεγονός ότι η χώρα σας αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου. Ότι η Κροατία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λετωνία στην Ευρωζώνη. Όλη η Ευρώπη θα μπορούσε να γιορτάζει αλλά δεν πάβει να αυξάνεται και ο αριθμό των ευρωσκεπτικιστών. Και δεν ξέρουμε και πώ αντιμετωπίζει όλε αυτέ τι εξελίξει η Ρωσία. Είμαι σίγουρο ότι τα έχουν καταγράψει πάντω προσεκτικά. Πάντω με εντυπωσίασε η ειλικρίνεια και το άνοιχτο σα πνεύμα. Το πρωί μου σε συνεδρίαση τη Επιτροπή Πολιτισμού, όπου ο Υπουργό σα και πάλι παρουσίασε τι προτεραιότητε του εξαμήνου τη Προεδρία σα. Αυτό που προέκυψε την Ατλαντική Προεδρία είναι ότι κάποιες φορέ νομίζω συζητούμε για κονδύλια, για χρήματα, περιμένουμε πολλά από τις προεδρίες. Ιδίω από μικρέ χώρε όπω η δική σα, σα φορτώνουμε πολλέ ευθύνε. Έχετε αναλάβει για πρώτη φορά την Προεδρία, άλλωστε. Αλλά εδώ είμαστε κι εμεί για να σα βοηθήσουμε, να σα στηρίξουμε. Ω προ τι προσδοκίε μα, λοιπόν. Στο δεύτερο εξάμεινο του 2013. Τι σκοπεύετε να κάνετε, γιατί κάποια πράγματα έχουν ήδη καθοριστεί από το πρώτο εξάμεινο της χρονιάς. Σίγουρα έχετε δύσκολες αποφάσεις να λάβετε. Αναφέρον οι συνάδελφοι την ε, πολλαπλή ερεσιμότητα, το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, τη συγχρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Ελπίζω ότι θα καταλήξετε όσο το δυνατόν περισσότερα αποτελέσματα, αλλά φοβάμαι ότι όταν ξεκινήσει η επόμενη χρονιά και θα αναλάβει η Ελλάδα, θα έχουμε ήδη περάσει σε αριθμό εκλογών. Θα επικεντρώνονται όλοι λιγότερο σε τέτοια ζητήματα που θα μας δυσκολεύουν κιόλας. Άρα αναλαμβάνεται σε μια καθοριστική περίοδο και για το τρίο προεδριών, την τρόικα προεδριών όπως έχει ονομαστεί. Ήθελα να ρωτήσω, δεν πιστεύετε ότι υπάρχει μια επικάλυψη στις προσπάθειες. Υπάρχουν μάλλον πολλοί εμπειρογνώμονες ταυτόχρονα, συμβάλλουν στον ίδιο σκοπό. Αυτό πώς το αξιοποιείτε, γιατί θέλω να με βέβαιος ότι θα κάνατε πολύ καλή δουλειά αλλά ας ε, θυμηθούμε τον εμπειρογνώμονα που μίλησε για το ρόλο των γυναικών και το πόσο καλή ισότητα, ισορροπία έχετε πετύχει εσείς ε, στην εκπροσώπηση των γυναικών. Ελπίζουμε αυτό να δώσει το παράδειγμα και να εξασφαλίσουμε συνέχεια στο έργο των Προεδριών. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι θα κάνατε πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε ο κύριος Συμπράσος. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πολύ που είστε παρόν. Ως εκπρόσωπος της ε, Λουθουανίας, με τέτοια ενεργητικότητα, σας εύχομαι να έχετε όλη την απαραίτητη ενεργητικότητα που θα χρειαστείτε για το εξάμεινο της Προεδρίας σας. Σας άκουσα να αναφέρεστε επανειλημμένα στην έννοια της προστιθέμενης αξίας. Ξέρουμε πολύ καλά και στη Λιθουανία και σε άλλα από τα πιο πρόσφατα κράτη-μέλη ότι η ανεργία αυξάνεται, η ανεργία των νέων αυξάνεται, υπάρχει ε, έξοδος από τη χώρα και οι πιστώσεις που θα έπρεπε να αξιοποιηθούν για να βοηθήσουν την οικονομική ανάπτυξη πολλές φορές πηγαίνουν για να ε, φτιάξουμε ακόμη περισσότερους δρόμους ε, στους οποίους ε, ταξιδεύουν πολύ λίγα αυτοκίνητα και για πολύ φαρδιά πεζοδρόμια που δεν έχουν λόγω της μετανάστευσης αρκετούς πεζούς για να βαδίζουν σε αυτά. Ε, πώς λοιπόν θα βελτιώσετε την κατάσταση. Τα συζητάμε πολλές φορές αλλά όταν πρέπει να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο υπάρχει μεγάλη αδράνεια. Ε, προκρίνουμε τα προγράμματα που μπορεί να είναι ευχερέστερο να εφαρμοστούν αλλά που δεν παρέχουν κατά ανάγκη προς τη θέμα αξία. Και περιμένω την απάντησή σας επειδή έχετε μεγάλη πείρα σε αυτό το τομέα. Μαρία Ριγόγεν. Ευχαριστώ. Παρακαλώ εδώ. Συμφωνώ ε, σε γενικές γραμμές με την παρουσίαση που κάνετε για τις ε, προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Ελπίζω να δώσετε την αναγκαία όθηση για να ε, αποκτήσει το ευρωπαϊκό όραμα και πάλι δυναμισμό. Θα ήθελα περισσότερη πληροφόρηση για αυτό που είπατε για την αναθεώρηση όλων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών γιατί ίσως μερικές να μην έχουν επαρκή προστιθέμενη αξία. Είπατε, θέλουμε να αλλάξουμε το κέντρο βάρους. Ξέρουμε ποιε ήσαν οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές, μία από τις μεγάλες επιτυχίες της ε, πολιτικής συνοχής. Γι' αυτό θα ήθελα περισσότερη πληροφόρηση. Άλλη μια φορά σας εύχομαι επιτυχή Προεδρία του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. ο Προεδρεύων. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Πριν απαντήσω στις επιμέρους ερωτήσεις, σαν σε διαβεβαιώ ότι η συνεργασία που είχαμε με την προηγούμενη Προεδρία, την Ιρλανδική, ήταν άριστη Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τις ε, προσωπικές επαφές που είχαμε. Ε, αυτό μας επιτρέπει να μοιραστούμε εμπειρίες, αλλά και να λάβουμε τις διαβεβαιώσεις των Ιρλανδών συναδέλφων. Ότι παρά το ότι έληξε η Προεδρία τους, είναι πάντα στη διάθεσή μας για να μας παράσχουν βοήθεια. Έχουμε κάποιον στο Υπουργείο Οικονομίας μας, που εργαζόταν για το στο Ιρλανδικό Υπουργείο Οικονομίας και επανήλθε και έτσι μπορεί να μας βοηθήσει. Αυτή η βοήθεια είναι απόλυτα αναγκαία. Ιδιαίτερα για χώρες σαν τη δική μου που είναι μικρή, αλλά και η Ιρλανδία είναι μικρή χώρα. Αλλά βέβαια η διαφορά είναι ότι είναι η πρώτη μας προεδρία ενώ εσάς ήταν η έβδομη. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που συζητήσαμε και με τον Υπουργό Νούναν και τους άλλους συναδέλφους του. Τι προσφέρει μια τεράστια εμπειρία προεδριών και ποια διαφορά από εμάς που είμαστε στην πρώτη μας. Και τελικά καταλήξαμε πως ε, δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Γιατί ε, μεταβάλλεται τόσο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση που κάθε φορά είναι σαν καινούργια. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε φάση τεραστίων αλλαγών και με πολύ ταχύ ρυθμό. Αυτό ίσως να μην αφορά τόσο πολύ τα θέματα περιφερειακής πολιτικής, αλλά για θέματα οικονομικής πολιτικής, για το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ, το οποίο έχω του οποίου έχω την τιμή να προεδρεύω. Είναι σαφές ότι για πολύ περίπλοκα θέματα όπως η Τραπεζική Ένωση η κατάσταση μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη και από τον σκεπτικισμό μέχρι την επίτευξη την ε, συζήτηση για το ποια λύση είναι η καλύτερη βλέπουμε απόψεις να αλλάζουν αντιδιαμετρικά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνέχεια μεταξύ Προεδριών. Εγώ ως μελλοντικός Προεδρεύων ήδη από τον ε, Ιανουάριο άρχισα να προετοιμάζομαι. Ήδη αρχές Δεκεμβρίου μετά τις εκλογές ανέλαβα αρμοδιότητες. Νομίζω ότι έκανα καλά που προετοιμάστηκα νωρίς και επίσης οι συνεργάτες μου είχαν πολύ συχνές επαφές με τους συναδέλφους από άλλα κράτη-μέλη, αλλά και με εσά και μέλη του προσωπικού σας. Είναι πολύ σημαντικό και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία και φυσικά ε, όλα τα ντοσιέ, όλη μας την εμπειρία ε, πιστεύω ότι με πολύ ομαλό τρόπο θα τα περάσουμε και στην Προεδρία την ελληνική. Φυσικά ε, όλοι είναι πάντα πολύ απαιτητικοί και οι πόροι και το προσωπικό είναι πάντα περιορισμένοι. Γι' αυτό σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη ότι και εσείς έχετε προεκλογική περίοδο, άρα και οι δικοί σας πόροι θα είναι περιορισμένοι, οι δικές σας δυνατότητες. Άρα θα πρέπει να επιδιώξουμε να συντονίσουμε τα προγράμματα εργασιών μας για να μην, έχουμε, ε, να μην χρειάζεται να περνάει υπερβολικά πολύς ε, χρόνος μέχρι να καταλήξουμε ε, σε αποφάσεις κάθε ουδέν καλό να μηγες κακού και αντίστροφα. Τώρα συγκεκριμένες ερωτήσεις. Λοιπόν, να απαντήσω στον Λιθουανό συνάδελφο και θα μιλήσω λιθουανικά. Αγαπητέ Γιώζας, έθεσες ένα ε, θεμελιώδες ερώτημα το οποίο προσπάθησα να αντιμετωπίσω και εγώ στην αρχική μου εισαγωγή αλλά και απαντώντας σε προηγούμενες ερωτήσεις. Φυσικά η εθνική αλλά και η ευρωπαϊκή πόρη είναι περιορισμένη Άρα πρέπει να βρούμε ευφυείς τρόπους ε, βελτιστοποίησης της χρήσης των πόρων. Και πιο αποτελεσματικής φυσικά. Νομίζω ότι ήδη ε, οι δέσμοι ε, μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δηλαδή, που αναφέρει αναλυτικά πώς πρέπει να δοθεί, να αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή στήριξη και στις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο συζητάμε νέες μεθόδους, νέους κανονισμούς ε, κατά την ε, περίοδο του νέου πολιετούς πλαισίου όπου θα έχουμε σε αυτό το κουτί με εργαλεία όπως το λέμε ακόμη περισσότερες δυνατότητε. και για την πολιτική συνοχής θα δοθούν λοιπόν νέες ευκαιρίες με βάση και τα αποτελέσματα και την κριτική αξιοποίηση των ε, αποτελεσμάτων της δουλειάς μας μέχρι τώρα και την πείρα των κρατών μελών που είναι στη διάθεσή μας. Όλα αυτά θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε. Γιάννα, θέσατε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα επιδιώξω λοιπόν και εγώ να είμαι ακριβής. Προσβλέπουμε σε πολιτικές συμφωνίες Σε αυτή την πορεία ε, είναι γενικά αρνητικό να θέτουμε καταληκτικές ημερομηνίε. Ότι μέχρι τότε πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Αλλά υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία. Είναι η πρώτη πρώτου 14. Αυτή είναι η προθεσμία. Οπότε, εάν δεν τηρηθεί, θα αποφασίσουν οι εκλογείς. Εάν είναι αποτελεσματική εάν βοηθάει τους πολίτες της η Ένωση ή όχι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι είναι ακόμη ζωντανή η Ευρώπη, γιατί πιστεύω ότι είναι ακόμη ζωντανή. Αλλά πρέπει να το αποδείξουμε με τις προσπάθειές μας. Η επίτευξη συμφωνίας σημαίνει ότι πρέπει να θέσουμε κατά μέρος κάποιες επιθυμίες, ε, φιλοδοξίες, απόψεις που μπορεί να είναι πολύ καλά όλα αυτά, για να επιτύχουμε συμφωνία εδώ και τώρα. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχετε πολύ επικοδομητική αντιμετώπιση. Οι συνεργάτες μου θα εργαστούν χωρίς διακοπές. Τις έχουμε ξεχάσει ήδη φέτος, τις διακοπές μας. Έχουμε σοβαρές προκλήσεις ενώπιόν μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δείξουμε ότι όντως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί συμφωνία. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε αποτελέσματα για τις πολιτικές προοπτικές και τον κανονισμό ή τους κανονισμούς της πολιτικής συνοχής. Η κανονική σειρά θα ήταν πολιτική συνοχής και μετά πολιετής ε, προοπτικές εν ώψη και των ε, πολιτικών συνθήκων. Από μεθοδολογικής απόψεως θα ήθελα ήδη να έχουμε τις πολιτικές προοπτικές επιτάπητους. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να εργαστούμε περισσότερο. Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος. Για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Η γενική προσέγγιση θα μας δοθεί μέχρι τέλος Ιουλίου από το Συμβούλιο, άρα θα μπορέσουμε, πιστεύω, να καταλήξουμε σύντομα. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι... Α, μα, μισό λεπτό. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές... Με συγχωρείς Μαρία! Βεβαίω, σε ορισμένε περιπτώσει σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Αλλά να παραδεχθούμε ότι ορισμένες φορές δεν ήταν και τόσο αποτελεσματικές αυτές οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές και χρειάστηκε να αξιοποιήσουμε άλλα μέσα περιφερειακής πολιτικής. Τώρα, καθαρά η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα πρέπει να έχουμε υπερβολικά μέσα σε κάθε τομέα πολιτικής. Ίσως λιγότερα μέσα που να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά να είναι καλύτερο. Δεν χρειάζεται να κατακαιρματίζουμε τους πόρους μας, όχι μόνο τους ε, οικονομικούς αλλά και τους ανθρώπινους πόρους. Πολλά μέσα όπου κανείς δεν έχει συνολική εικόνα. Αυτό βέβαια δεν αφορά την ε, μακροπεριφερειακή στρατηγική. Θα εξακολουθήσει να είναι ε, σημαντικό μέσο πολιτικής. Ήδη ε, έχουμε αξιοποιήσει αυτό το μέσο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για μας βέβαια η, περίοδος της Βαλτικής, η περιοχή της Βαλτικής και η μακροπεριφερειακή στρατηγική σε αυτήν την περιοχή είναι πολύ σημαντική και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναθεώρησης που έχει συμφωνηθεί εδώ και πολύ καιρό θα αναθεωρηθεί κατά το τρέχον εξάμεινο. Και χαίρομαι που συμπίπτει με την Λιθουανική Προεδρία. Δεν θα επιδιώξουμε να ασκήσουμε υπερβολική επιρροή, όχι βέβαια. Αλλά κάτι τέτοιες συμπτώσεις ε, συμβαίνουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτιμώντας την ε, μακροπεριφερειακή στρατηγική στη Βαλτική δεν θα εξαγάγουμε συμπεράσματα γενικότερα για αυτή τη στρατηγική. Γιατί πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα και από τα θετικά αλλά και να τονίσουμε και να εξαγάγουμε πορίσματα και από τις αποτυχίες, τα αρνητικά για να εξετάσουμε τις βελτιώσεις που χρειάζονται. Τώρα νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε, που μοιραστήκατε μαζί μας τις ανησυχίες σας και τις φιλοδοξίες σας και όντως τέλη Αυγούστου θα έχουμε ήδη τη συνάντηση. Ξέρω ότι το προσωπικό μας θα φροντίσει έτσι κι αλλιώς αύριο το πρωί θα συναντηθούμε με τον Ντάριους και την Κριστίν για το τελευταίο τριμερή διάλογο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ελπίζουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε πλήρως τις ευκαιρίες που θα έχουμε το Σεπτέμβριο για να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες και έτσι στη δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου να έχουμε παρατέρω αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πάντως που θα αναλάβετε τη διαμεσολάβηση και θα βοηθήσετε να προχωρήσει η διαδικασία και στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν και όλες μας τις ευχές για Καρποφόρα Προεδρία. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε, μην ε, φύγετε από την αίθουσα. Uh, θα έχουμε το δικό σας σημείο, το σημείο 16 στην ημερήσια διάταξη, έτσι. Παρακαλώ κύριε Μπράσας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ για να συμμετάσχετε σε αυτήν την πρώτη συζήτηση όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης για την ηλεκτρονική υγεία για την περίοδο 2012-2020. Πρέπει να στηρίξουμε, πιστεύω, την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί η ηλεκτρονική υγεία. Είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να χρησιμοποιήσουμε την πληροφορική. Και μπορεί μάλιστα να βοηθήσει ακόμα περισσότερο με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί υγεία. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε τρεις πτυχές. Πρώτα απ' όλα το θέμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Μέσω της ηλεκτρονικής υγείας βελτιώνεται. Το πρόγραμμα αυτό δράσης προσφέρει νέες ευκαιρίες, νέες δυνατότητες. Άρα η πρόσβαση αυτή θα είναι πιο εύκολη και για περισσότερο κόσμο. υπάρχουν πολίτες ε, οι οποίοι λόγω οικονομικής κατάστασης, κοινωνικής ηλικία δυσκολεύονται σήμερα. Ε, αυτοί θα διευκολυθούν. Δεύτερον, προκειμένου οι υπηρεσίε ε, υγείας να είναι εύκολα προσβάσιμες στον κόσμο, πρέπει να καταρτήσουμε τους ασθενείς για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική υγεία τους ασθενείς αλλά και τους επαγγελματίες του κλάδου. Άρα πρέπει να μάθουν να χειρίζονται την πληροφορική. Και εδώ είναι που τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν ε, μεγάλες προσπάθειες, ευρυζωνικότητα για παράδειγμα. Οι περιφερειακές, οι τοπικές αρχές έχουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατί βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη. Θα ήθελα επίσης να πω ότι χαίρομαι πολύ ότι από τη μέχρι τώρα εμπειρία βλέπουμε ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί και πολλές έχουν υιοθετήσει προγράμματα ηλεκτρονικής υγείας. Ενθαρρύνουμε λοιπόν τις αρχές αυτές προκειμένου να χρηματοδοτήσουν ακόμα περισσότερο τέτοια προγράμματα ηλεκτρονικής υγείας και να φροντίσουν να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και περιμένω τώρα να ακούσω τι προτάσεις έχετε εσείς, τι τροπολογίες θέλετε να προτείνετε. Πιστεύω ότι με καλή συνεργασία μεταξύ μας θα βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Οι σκιώδες δεν είναι στην αίθουσα. Μήπως κάποιος εκ μέρους τους θέλει να πάρει το λόγο. Νίκο, εσείς είσαστε σκιώδες ή όχι. Μια που είσαστε εδώ. Σας έχουμε στον κατάλογο. Ε, πράγματι οι υπηρεσίες ε, e-health είναι σημαντικές γιατί σήμερα εξαιτία της κρίσης έχει, έχουν υποβαθμιστεί πολλές υπηρεσίες υγείας ήδη σε περιοχές που ήταν απομακρυσμένες ε, υπήρχαν ορεινές περιοχές, υπήρχαν ισιωτικές περιοχές υπήρχε πρόβλημα πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. σήμερα αυτό έχει επιδεινωθεί ειδικά στις χώρες της κρίσης του Νότου ε, υπάρχει μια αποδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας τουλάχιστον στο βαθμό που ε, έχω την εικόνα αυτή από την Ελλάδα και από άλλες περιοχές υπάρχουν μείωση του προσωπικού, υπάρχουν υπηρεσίες που κλείνουν και αυτή τη στιγμή οι πολίτες είναι διπλά επιβαρημένοι. Απ' τη μια μειώνεται το εισόδημά τους και απ' την άλλη έχουν περιορισμένη πρόσβαση υπηρεσίες υγείας κατά καιρού έχουν στηθεί τα θέματα της ε, πρόσβαση μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην υγεία, κάτι το οποίο θα διευκόλυνε ιδιαίτερα ε, του ανθρώπου που βρίσκονται σε μικρά νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αρκεί να βρεθούν όμως και κατάλληλα εργαλεία να στηρίξουν τέτοιες ε, παρεμβάσεις και τέτοιες επενδύσεις. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στα θέματα της κοινωνικής συνοχής, να μειωθεί δηλαδή η σε απομακρυσμενες περιοχες και νομιζω οτι ειναι κατι παρα πολυ σημαντικο αρκει να βρεθουν ομω και καταλληλα εργαλεια να στηριξουν τετοιε παρεμβασει και τετοιε επενδυσει νομιζω οτι θα βοηθησει παρα πολυ στα θεματα της κοινωνικης συνοχης να μειωθει δηλαδη η ε, αυτές οι ανισότητες που μεγενθύνονται σήμερα στην πραγματικότητα. Δηλαδή θεωρούμε ότι ο πολίτης σε κάθε περίπτωση δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσία υγείας. Και αντίθετα βλέπουμε σήμερα ότι στοιχειώδεις τέτοιες υπηρεσίες για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στερούνται και όχι μόνο ε, για αυτούς που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά και αυτούς που είναι σε πόλεις. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβαση μέσα από τη χρήση και τεχνολογίας πληροφορικής. Κατά καιρούς έχουν δοκιμαστεί τέτοια συστήματα, σε ορισμένες χώρες έχουν καλή εφαρμογή. Νομίζω όμως ότι αυτές που χρειάζονται περισσότερο τέτοιες υπηρεσίες είναι οι χώρες που, δεν, που έχουν σήμερα, βιώνουν σήμερα την κρίση. Ε, μπορούμε να καταθέσουμε προτάσεις πιστεύω και ιδέες για να μπορέσουν να επιταχυνθούν τέτοιες παρεμβάσεις σε αυτές τις περιοχές. Ε, είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και αναγκαίο στη σημερινή συγκυρία. Thank Σας ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει άλλος σκιώδης εδώ. Α, παρακαλώ, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε εποφελούμε από την ευκαιρία αυτή, γιατί στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την ηλεκτρονική υγεία και θα ήθελα να σας αναφέρω εδώ κάποιες σκέψεις της εισηγήτριας. Όσον αφορά την γύρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη. Όντως θα πρέπει να προχωρήσουμε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Η υγεία είναι πολύ βασικός πυλώνας του κράτους ευημερία και γι' αυτό και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η πληροφορική και η εφαρμοσμένη επικοινωνία ώστε να τις χρησιμοποιήσουμε και στην υγεία. Γιατί έτσι θα εκδημοκρατήσουμε την υγεία. Θα φτάσει η υγεία εκεί όπου δεν έφτανε μέχρι τώρα και θα εξυπηρετήσει τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν πάντα την ευκαιρία να πάνε να δουν έναν καλό ειδικό γιατρό. Θα μπορέσουν να συνδεθούν όμως μέσω της πληροφορικής ε, πια. Η ηλεκτρονική λοιπόν υγεία μπορεί να βοηθήσει και την ποιότητα της ζωής των ηλικιωμένων. Όμως πρέπει να επενδύσουμε προηγουμένως, να επενδύσουμε στα στοιχεία εκείνα που δεν είναι γνωστά στους ηλικιωμένους ή και γενικότερα στους ασθενείς και πολλές φορές δεν τα γνωρίζουν ούτε καν ήδη οι επαγγελματίες του κλάδου, το προσωπικό δηλαδή υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, αν δεν υπάρχει κανείς άλλος που θέλει το λόγο, να προσθέσω εγώ κάτι. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής 2000 με 2006 έχει επενδύσει στις ε, υπηρεσίες αυτές υγείας με διάφορα προγράμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπορούμε λοιπόν να χτίσουμε πάνω σε αυτά, να αποφεληθούμε δηλαδή από αυτές τις εμπειρίες και να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει να αποφασίσουμε προθεσμία για υποβολή τροπολογιών προτείνονται 12 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στη γνωμοδότηση του κύριου Βίνκλερ. Είναι το σημείο 22. Πρόκειται για τις στρατηγικές εφιούς εξειδίκευσης. Παρακαλώ κύριε Βίνκλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η στρατηγική για την ευφυή εξειδίκευση είναι στην ημέρηση διάταξη. Οι περιφέρειε θα πρέπει να έχουν μια περιφερειακή στρατηγική για τι επενδύσει, την έρευνα και την καινοτομία με τη νέα μέθοδο τη ευφυού ε, εξειδίκευση. Εάν θέλουν να λάβουν χρηματοδότηση για το θεματικό στόχο 1, έρευνα και καινοτομία εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις ε, εάν δεν έχει η Κομισιόν λάβει την εξάντε αιρεσιμότητα θα διακόπτει την χρηματοδότηση. Επειδή βέβαια έχουμε ύφεση αυτή τη στιγμή, θα μας βοηθούσε αυτό να αξιοποιήσουμε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για να προχωρήσει η Ένωση της Καινοτομίας και η Ένωση να γίνει πιο καινοτόμα και άρα πιο ανταγωνιστική. Η χρονική στιγμή που συζητάμε την έκθεση δεν είναι βέβαια ιδανική. Οι διαπραγματεύσει για το νομοθετικό πλαίσιο για τα διευθυντικά ταμεία κλείνει αυτή τη βδομάδα. Οι περιφέρειες ε, ε, έχουν διαφορετικό ε, βαθμό εξειδίκευση τη στρατηγική τους και οπωσδήποτε πρέπει οι περιφέρειες να συντονίσουν τα προγράμματά τους με τα προγράμματα γενικότερα καινοτομίας και επενδύσεως. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ρέγγιο ξέρουν τι γίνεται στις διάφορες περιφέρειες, άρα θα ήταν καλό να γίνει ένας πρώτος ενδιάμεσο απολογισμός ποιες προκλήσεις μπορούν να βοηθήσουν άλλοι ε, παράγοντες της ε, περιφέρειες να αντιμετωπίσουν έχοντας ακούσει από διάφορους εμπλεκομένους μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και ίσως να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στο μέλλον. Ως βάση της πρώτης ανταλλαγής απόψεων έχετε λάβει το έγγραφο εργασίας που εξεπώνησα. Πρέπει να δούμε ευρύτερα τα θέματα και θέτω μερικά κρίσιμα ερωτήματα, πιστεύω, η Κομισιόν και εμείς πρόσφατα καταλήξαμε σε ε, έναν ορισμό το τι σημαίνει αυτή η στρατηγική αλλά να σας πω εγώ με τα δικά μου λόγια περί τίνος πρόκειται. Κάθε περιφέρεια θα πρέπει μαζί με τους εταίρους της την έρευνα και την καινοτομία και ιδιαίτερα με τις επιχειρήσεις να αναλύσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της και να δημιουργήσει τη δική της προοπτική με λίγες προτεραιότητες πώς θα μπορούσαν να ενισχύσουν την καινοτομία τους οι περιφέρειες και άρα την ανταγωνιστικότητά τους και συνολικά την ανταγωνιστικότητά της Ένωσης. Ιδιαίτερο πρέπει να είναι το θέμα πώς θα αξιοποιήσουμε τις ε, ε χρηματοδοτήσεις για την έρευνα ε, και την καινοτομία και ιδιαίτερα στα πλαίσια του ορίζον 2020. Ιδεοδός οι περιφέρειες θα πρέπει να συμπληρώνονται. Να θέσω τα σημαντικότερα θέματα που με απασχόλησαν για να βοηθήσω την ανταλλαγή απόψεων. Πρώτον, η εξάντε ερεσιμότητα δεν ε, Υπάρχει κίνδυνος να είναι μια καθαρά τυπική διαδικασία. Οι περιφέρειες μπορούν να δημιουργήσουν μια προοπτική και η Κομισιόν απλώς εξετάζει τη μέθοδο. Αν υπάρχει δηλαδή γενικά μια στρατηγική και αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής στρατηγικής. Οπότε υπάρχει κάποιος κίνδυνος ότι μόνο τα πιο απαραίτητα θα γίνονται. Πρέπει να είναι σαφές ότι αυτή η εξάντε αιρεσιμότητα δεν είναι βέβαια και πανάκια. Η εφαρμογή θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική και δαπανηρή για τις περιφέρειες και αν οι περιφέρειες δεν καταλάβουν ότι είναι προς το συμφέρον τους η εκπόνηση μιας τέτοιας στρατηγικής και αν θεωρήσουν ότι είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, τότε δεν θα επιτύχουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να είναι αυτό σπυρούνισμα για να κάνουν οι περιφέρειες πράγματα που δεν έχουν κάνει πολύ μέχρι τώρα. Δεύτερον, αποφασιστικό ερώτημα. Μπορεί αυτή η στρατηγική να είναι η επιτυχής αντίληψη για όλες τις περιφέρειες, ανεξάρτητα πόσο αναπτυγμένες είναι, πόσο πολύ ενδιαφέρονται για την ε, καινοτομία. Γιατί ξέρετε πως είναι διαφορετικό το επίπεδο ανάπτυξης και διαφορετικό το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των ε, διαφόρων εμπλεκομένων και διαφορετική και η διοικητική υποδομή. Άρα πρέπει να προσαρμοστεί και η στρατηγική. Με ένα copy-paste δεν κάνουμε τίποτα. Δεν θα λειτουργήσει μια αντιγραφή τη στρατηγική μια άλλη περιφέρεια. Πρέπει να γίνει μια αρχική ανάλυση. Δεν μπορεί κάθε περιφέρεια, για παράδειγμα, να είναι ηγετική σε τεχνολογίε κλειδιά. Πρέπει να υπάρχουν περιφέρειε που θα αξιοποιήσουν την πείρα τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν αλλού. Καινοτόμω δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι εμεί είμαστε στου τομεί ψηλή τεχνολογία και μη τεχνολογική καινοτομία είναι πολύ ενδιαφέρον ε, ε, για παράδειγμα στον τομέα των υπηρεσιών, ε, στο δημογραφικό τομέα, σε κοινωνικά θέματα, στην υγεία. Δεν μπορούν όλες οι περιφέρειες να κάνουμε τα πάντα. Αυτή η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης τι είναι, είναι μια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω που βοηθάει να συμμετάσχουν οι εμπλεκόμενοι. Έτσι θα βοηθήσουμε να ενδιαφερθούν οι επιχειρήσεις, να καταλάβουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και προτερήματά τους, ποιο είναι το όραμά τους για το μέλλον. Η επιστήμη και η Κομισιόν πάντα είναι υπέρ αυτής της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω. Bottom up και όχι top down. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε προσεκτικά. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και οι άνθρωποι που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Και φυσικά ε, δεν θα είναι ικανοποιημένοι όλοι οι φορείς με τις αποφάσεις. Αλλά η ιδέα είναι σωστά. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος όπου δεν ακούγαμε αρκετά, δεν, αρκετά, δεν συνδυάζαμε αρκετά στη δουλειά μας τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Όλα αυτά ε, ακούγονται ωραία θεωρητικά, πρακτικά η εφαρμογή τους θα είναι πιο δυσχερής. Σε διάφορες περιοχές άκουσα να μου λένε ότι δεν μας ρωτάνε αρκετά, ότι συνεχίζουν να κάνουν αυτά που έκανε και παλιότερα. Έτσι όμως δεν γίνεται μια ουσιώδης ε, αυτοανάλυση. Πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας και των υπηρεσιών. Πρέπει οι υπηρεσίες να έχουν ένα πιο ευέλικτο τρόπο δράσης και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. Στις περιφέρειες, όπου η διοίκηση συνδυάζεται με τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τους επιστήμονες, τότε σε αυτές τις περιφέρειες έχουμε καλύτερες ε, πιθανότητες επιτυχίας. Και το νευραλγικό είναι η συμμετοχή των επιχειρήσεων. Ο χρονικός ορίζον για εκπόνηση αυτής της στρατηγικής είναι ρεαλιστικός. Πολύ σημαντικό σημείο. Για να έχουμε σύντομα νέες στρατηγικές και παρόλα αυτά να γίνει θεμελιώδης ε, κριτική αυτοανάλυση και για να ε, ρωτήσουμε και παρκώς τους εμπλεκόμενους φορείς ε, είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αν η εξάντε ρεσιμότητα έχει πληρωθεί. Πρέπει λοιπόν οι περιφέρειες να μπορούν να υποβάλουν και εναλλακτικά προγράμματα στρατηγικής που να περιέχουν και χρονοδιαγράμματα. Η εξάντε αιρεσιμότητα θα πρέπει το αργότερο μέχρι τέλους του 2016 να έχει ελεγχθεί και μετά η Κομισιόν θα πρέπει να εξακολουθεί να επιτηρεί προσεκτικά. Σε πολλούς τομείς όμως οι περιφέρειες έχουν ήδη καταρτήσει στρατηγική καινοτομία και ε, ορισμένοι έχουν ε, δεκαετίες εργαστεί για τέτοιες στρατηγικές. Αυτό καταδεικνύει ότι η κατάρτιση μιας τέτοια στρατηγικής είναι μακροχρόνια διαδικασία που θέλει επαρκή χρόνο. Από την άλλη μεριά πρέπει να φροντίσουμε να μην γίνει ανακύκλωση παλαιών στρατηγικών, να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Η νέα αυτή στρατηγική δεν πρέπει να οδηγηθεί ad absurdum. Πώς θα θέσουμε τώρα τις σωστές προτεραιότητες. Πολλές ε, περιφέρειες θέτουν ε, πολλές προτεραιότητες, ε, τις βάζουν παραθετικά και γι' αυτό επειδή είναι δύσκολη η οικονομική κατάσταση ε, ποντάρει κανείς σε πολλά άλογα. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα μπορέσουμε να κάνουμε την αναγκαία συγκέντρωση προσπαθειών. Ούτως ή άλλως όμως το σημαντικό είναι ε, να καταλάβουμε ότι όσο πιο ειδικευμένη είναι μια προσπάθεια τόσο μεγαλύτερο είναι ο κίνδυνος για την ε, ε, περιφέρεια. Αλλά από την άλλη μεριά η ευρεία προώθηση πολλών τομέων λόγω των οικονομικών δυσχεριών δεν είναι δυνατή. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ακριβώς ευφυή εξειδίκευση. Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε διαδικασίες που να είναι ήδη συγγενή με ορισμένα υπάρχοντα. Αυτό λέγεται ε, συγγενής ανάπτυξη. Μια τέτοια ευφυής ανάπτυξη που βοηθάει επίσης ε, ε, εάν συνδυάζει τις ίδιες διαδικασίες και τα ίδια προϊόντα σε πολλούς τομείς. Κατά τη γνώμη μου, οι περιφερειακοί παράγοντες είναι πολύ βασικό να εμπλακούν από νωρίς γιατί έτσι μειώνουμε τον κίνδυνο να μην επιτύχουμε στο τέλος. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να βελτιωθεί αυτή η συμμετοχή. Οι περιφέρειες πρέπει πάντα να έχουν δυνατότητα αλλά και το θάρρος να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους κατά την εφαρμογή εάν δεν λειτουργεί. Γι' αυτό χρειάζεται όχι μόνο σύστημα εποπτείας αλλά κάτι πολύ πιο έντονο. Τέλος, η εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργάνων της Ένωσης, ε, πώς θα μπορούσαν να, ε, η συνεργασία αυτή πώς θα μπορούσε να γίνει, πρέπει να το σκεφτούμε. Πώς οι πιστώσεις ε, σε αυτό το τομέα μπορούν να συνδυαστούν με άλλες χρηματοδοτήσεις από άλλα προγράμματα ή με ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις. Προσπαθούμε για παράδειγμα να συνδυάσουμε την χρηματοδότηση της έρευνας με την ε, χρηματοδότηση της συνοχής εδώ και δεκαετίες χωρίς να το επιτυχάνουμε. Πρέπει να το επιτύχουμε. Πρέπει λοιπόν στις ε, περιφέρειες να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις χρηματοδοτήσεις για την έρευνα και την ε, καινοτομία. Θα θέλαμε να συμμετέχουμε περισσότερο λοιπόν στις προτεραιότητες του 2020. Πρέπει να υπάρξει ευρύτερη συμμετοχή και να συμμετάσχουν και οι πιο ανεπτυγμένες περιοχές και οι περιφέρειες που δεν μπορούν να επιτύχουν αυτήν την ε, θαυμάσια καινοτομία πρέπει να συμμετάσχουν και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χέρμαν, λίγο πιο αργά, λίγο πιο αργά. Δύο λεπτά λέει ο κύριος Βίνκλερ. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει περισσότερη εκπόνηση λεπτομεριών να εκπονήσουμε το νομικό πλαίσιο. Είναι τόσο ε, δυσχερής η προσπάθεια προσαρμογής που είμαι κάπως ε, διστακτικός. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα τόσο στην εισαγωγή γιατί πιστεύω ότι αυτό θα διευκολύνει την περαιτέρω συζήτηση. Τίθεται το ερώτημα. Οι περιφέρειες έχουν επαρκή ε, ε, πλαισίωση στις προσπαθίες τους. Ποιοι, του δίνουν, ποιοι τους δίνουν σύμβολες. Πιο αργά να μιλάτε παρακαλώ λέει. Πιο αργά η πρόεδρος. Λοιπόν, τι συμβουλές, ποιοι συμβουλεύουν τις περιοχές που θέλουν να συμμετάσχουν και αυτές που πρέπει να συμμετάσχουν. Οι περιφέρειες έχουν στενή επαφή με την Επιτροπή ιδιαίτερα με τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο, η οποία είναι υπεύθυνη για την έγκριση των ε, προγραμμάτων και την ε, στρατηγική καινοτομίας. Άρα ε, και η χορήγηση συμβουλών και η έγκριση των προγραμμάτων γίνονται από τον ίδιο φορέα. Οπότε εδώ τίθεται το ερώτημα. Και επίσης Έχουμε και την εργασία της πλατφόρμας για την ΕΦΗ e, εξειδίκευση που έχει ε, συσταθεί στην Σεβίλη και που δίνει τη δυνατότητα μέσω εκτίμησης από ειδικού, αλλά έχουν κάνει αίτηση 130 περιφέρειες πολλές περιφέρειες θεωρούν ότι η συμμετοχή δεν θα τους δώσει ε, προστιθέμενη αξία, οπότε χρειάζεται ανάγκη ε, να βελτιωθεί η κατάσταση και να ενημερώσουμε καλύτερα διάφορες περιφέρειες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει περισσότερη επαφή και με άλλες γενικές διευθύνσεις όπως η Γενική Διεύθυνση Έρευνας. Τώρα η εξωτερική διάσταση των διαφόρων περιφερειών πώς θα διαμορφωθεί είναι ρεαλιστικό να την επιδιώξουμε οι ε, συνθήκες του πλαισίου είναι επαρκείς. Πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η πολιτική μας στον τομέα αυτό για όλες τις περιφέρειες. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμόσουν την εξωτερική διάσταση οι περιφέρειες. Δεν θα πρέπει να έχουν μια καλή στρατηγική για αυτές, αλλά να επιδιώκουν και συνεργασίες με άλλες περιφέρειες. Ιδεοδός, οι περιφέρειες θα έπρεπε να παίζουν συμπληρωματικό ρόλο. Αυτό ενισχύει και την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία σε όλη την Ένωση. Αλλά μόνο η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο έχει μια συνολική εικόνα της κατάστασης. Μόνο αυτή μπορεί να εισαγάγει κάτι τέτοιο. Όμως δεν μπορεί να παρέμβει η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο στον καθορισμό των ε, προτεραιοτήτων. Άρα θα πρέπει ε, να το κάνει αυτό κάθε περιφέρεια σε συνεννόηση με άλλους. Μεγάλη επιτυχία είναι η Silicon Ευρώπη που υπάρχει, αλλά μπορεί να απτυχθεί πολύ περαιτέρω η συνεργασία των περιφερειών στον τομέα αυτό. Η συνεργασία των περιφερειών βέβαια είναι περίπλοκη υπόθεση. Οι διαδικασίες προσαρμογής ακόμη και εντός μίας μόνο περιφέρειας είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Εάν επιχειρήσουμε να υπάρξει συντονισμός μεταξύ διαφόρων περιφερειών στα λειτουργικά προγράμματα, θα έχουμε μεγάλες δυσχέρειες. Στο μέλλον θα δούμε εάν είναι επαρκές το νομικό πλαίσιο. Εν πάση περιπτώσει, θα χρειαστεί ένας χρόνος για την αρχική εφαρμογή του προγράμματος για το, να μπορέσει το πρόγραμμα να λειτουργεί κανονικά. Θα χρειαστούμε πολύ χρόνο. Χρειάζεται φυσικά και συνεργασία ευρύτερων περιοχών αλλά αυτό θα σήμαινε μια ε, πολύ υψηλή χρηματοδότηση από ό,τι αποδέχονται οι κυβερνήσεις τώρα. Αλλά βεβαίως για ε, μεθοριακές περιοχές θα είχαμε μεγάλες εξοικονομίες στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει λοιπόν που βλέπω να υπάρχουν οι προκλήσεις. Προσβλέπω στη συζήτηση και στην Επιτροπή και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much. I would like to say that... Ευχαριστώ πολύ. Η γραμματεία δεν έχει λάβει από τους κοιόδης εισηγητές καμία ειδοποίηση. Αλλά το θέμα είναι θεμελιώδη σημασία. Ελπίζω λοιπόν να μα ενημερώσουμε, να μας ενημερώσουν ο κ. φανίσταλτοι. Λάμπερ. Ευχαριστώ, Πραγματικά το θέμα αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερο Είναι ένα πρώτο βήμα για να έχουμε το κείμενο ίδιας πρωτοβουλία που ε, επιδιώκουμε. Πολύ καλό το υλικό αυτό που μας παρουσιάσατε για να έχουμε μια πρώτη συζήτηση και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Διότι θα έχουμε τις πρώτες προτάσεις από τα κράτη-μέλη επιτάπητος στο πρώτο μέρος της επόμενης χρονιάς, στο πρώτο εξάμεινο. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα να λαμβάνονται υπόψη. Ε, για την ώρα έχουμε περισσότερε ερωτήσει και απορίε παρά απαντήσει. Και στρέφομαι και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και επισημένω τι προτάσει των κρατών που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στι συμφωνίε εταιρική σχέση. Ερώτηση λοιπόν προ τον κύριο Βίνκλερ, Πώ προγραμματίζεται να γίνουν όλα αυτά, διότι αν ψηφίσουμε στις αρχέ τη επόμενη χρονιά. Ίσως τις συγκεκριμένες πληροφορίες, τα δεδομένα να τα έχουμε στα χέρια μας. Και να έχουμε και μια πιο σαφή εικόνα για το τι πρόοδος έχει επιτελεστεί στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω και κατά δεύτερον χαίρομαι πολύ που έχετε μια διαλεκτική προσέγγιση ε, ανοιχτό μυαλί. Απλώς αυτό που μου έρχεται κατά νου είναι το αποδείξτε το, ε, δείξτε μας πώς γίνεται. Δεν ξέρω σε όλε τι ερωτήσει που έχετε θέσει ποιο μπορεί να απαντήσει. Κάποιε φορέ είναι λίγο ρητορικέ. Φαίνεται να απαντάτε μόνο σα. Ή μπορείτε να απαντήσετε εδώ, ίσω η Επιτροπή των Περιφερειών. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα και κάποιες παρατηρήσεις ε, να κάνω εδώ για να ληφθούν υπόψη. Υπάρχουν κάποια εργαλεία που θα μπορούσατε να τα συμπεριλάβετε. Τα αποτελέσματα λόγου χάρη της νομοθετικής μας πρότασης για το EIT, την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Τεχνολογία. Υπάρχουν και τα περιφερειακά προγράμματα καινοτομία που είναι παρόμοιοι τρόποι, παράλληλοι δρόμοι που θα μπορούσαν να καλύπτονται από αυτή τη στρατηγική εξειδίκευση στις περιφέρειες δηλαδή με καλλιέργεια της ε, καινοτομίας και της έρευνας μέσω του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Καινοτομία και την Έρευνα και την Τεχνολογία μάλλον. Πολλοί από τους τομείς αυτούς θα μπορούσαν να καλύπτονται εδώ και να κάνετε και τους κατάλληλους σχετισμούς. Έπειτα μιλήσατε για την εξωτερική διάσταση. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν εδώ ευρωπαϊκοί μηχανισμοί. Όπως με την Ευρωπαϊκή Υποδομή για την Έρευνα, το ΕΡΙ, όπως είναι γνωστό. Υπάρχει αυτό το εργαλείο, υπάρχει ο μηχανισμός και δίνει στις περιφέρειες, στα Ινστιτούτα του, στα Ιδρύματα Έρευνας και ε, καινοτομίας να λάβουν κάποιο καθεστώς, νομικό καθεστώς ε, μέσω και βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Γιατί κάποιες φορές μιλάμε για εξωτερική διάσταση και το ονομάζεται μαύρο κουτί, αλλά εκεί πρέπει να βοηθήσουμε να τους βοηθήσουμε να βρουν εταίρους και συνεργάτες στους τομείς ειδικευσής τους, είτε είναι αυτοκινητοβιομηχανία, είτε είναι τεχνολογία. Πολλές από τις δραστηριότητες τους μπορούν να διαρθωθούν έτσι, που να πάρουν διασυνοριακές διαστάσεις και να γίνουν ευρωπαϊκές. Σκεφτείτε και αυτή την οπτική γωνία. Επίσης, συμφωνώ ότι θα πρέπει να δώσουμε κάποια απόκριση και κάποια συνέχεια στις περιφέρειες της γνώσης. Δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση για την ερώτησή σας, εάν αυτό καλυπτόταν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ή όχι. Αλλά τώρα δεν ισχύει πια. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα Horizon, Horizon 2020. Γιατί, Γιατί η περιφερειακή πολιτική με αυτή τη νέα μορφή που έχει πάρει μπορεί να καλύπτει αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Θα γίνει όμως ή όχι. Ίσως ο εισηγητής να ξέρει να μας πει ή να το μελετήσει. Νομίζω πραγματικά όμως ότι έχετε θέσει πολλά εύστοχα ερωτήματα σε αυτή τη χρονική περίοδο και ίσως να μας έλεγε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις δικές της τις ε, απόψεις. Νομίζω είναι καλή στιγμή να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα ως Κοινοβούλιο, να δούμε τι θα προκύψει τους ερχόμενους μήνες. Ευχαριστούμε κύριος Χρυσόγελος. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, γιατί αν θέλουμε να βγούμε από αυτή την κρίση που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα στον Νότο, θα πρέπει να βασιστούμε στο θέμα της καινοτομίας σε καινούργιες ιδέες και σε καινούργιες ε, μορφές παραγωγής και αυτό προϋποθέτει πράγματι να περάσουμε από ένα μοντέλο ε, που ήταν συγκεντρωτικό στην έρευνα και τεχνολογία που γίνονταν κυρίως σε κρατικό επίπεδο πολλές φορές ή σε επίπεδο μεγάλων επιχειρήσεων να περάσουμε σε ένα πιο αποκεντρωμένο ε, μοντέλο παραγωγής έρευνας και τεχνολογίας. Ε, είναι, όταν μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη είναι απαραίτητο να ξέρουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας περιοχής, ποια είναι τα δυνατά της σημεία, ποιες είναι οι αδυναμίες και τι πρέπει να κάνουμε για να ξεπεράσουν αυτά εκεί που υπάρχουν ε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά να τονιστούν και οι αδυναμίες να αντιμετωπιστούν. Μιλώντας για τα νησιά παράδειγμα, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πολλές φορές θα αντιμετωπίζουμε ως προβλήματα, ως μειονεκτήματα, αλλά αν αλλάζαμε τον τρόπο προσέγγισης και υπήρχαν κατάλληλα εργαλεία, αυτά θα γίνουν πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, ένα νησί είναι ένα κλειστό οικοσύστημα. Η έρευνα λοιπόν εκεί για οικολογικές μορφές γεωργίας, ή για χρήση της βιο, ε, βιοοικονομίας είναι ε, πολύ ενδιαφέρουσα. Αν πράγματι όμως μπορέσουμε σε αυτά τα μέρη να αντιληφθούμε ότι εκεί είναι το μέλλον τους. Δηλαδή σε καινούργιες ιδέες, σε οικολογική καινοτομία, σε καινούργιες ιδέες. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι συνήθως αυτές οι περιοχές δεν έχουν δικιά τους έρευνα, δεν έχουν δικιά τους ε, αναζήτηση λύσεων, αναπαράγουν παλιά μοντέλα και εκεί έχουμε τώρα η κρίση επιδεινώνει ακόμα περισσότερο αυτή την απόσταση που υπάρχει μεταξύ περιοχών που έχουν την ικανότητα τα ερευνητικά κέντρα να προχωρούν σε έρευνα να μπορούν να αναπτύσσουν περιφερειακή στρατηγική έρευνας και τεχνολογίας και περιοχές οι οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν εντελώς στοιχειώδη θέματα και μάλιστα αναπαράγοντας παλιές λύσεις. Να ένα παράδειγμα. Ε, δεν ανάγκη να έχουμε πάντα το ίδιο μοντέλο επεξεργασία των λιμάτων, το οποίο είναι έργα πολιτικού μηχανικού, τσιμέντα κλπ. Προφανώ υπάρχουν πολύ διαφορετικέ λύσει για να επεξεργαστούμε τα λίματα ε, από οικισμού, από πώληση, από ξενοδοχεία κτλ. Αλλά ποιο θα κάνει αυτή την έρευνα στο περιφερειακό επίπεδο να βρει κατάλληλα συστήματα. Θα έρθει μια εταιρεία, θα προτείνει ένα μοντέλο, παραγωγή, ένα μοντέλο επεξεργασίας των λιμάτων και έτσι βλέπουμε πολλές φορές στην περιφερειακή πολιτική να χρηματοδοτούμε μέσα από το Ταμείο Συνοχής έργα τα οποία κοστίζουν 1,5 εκατομμύριο, τα οποία δεν λειτουργούν όμως γιατί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ε, του ανθρώπινου δυναμικού ή των ικανοτήτων που υπάρχουν σε μια περιοχή. Άλλες λύσεις θα ήταν κατάλληλα προσαρμοσμένες, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πολύ πιο οικονομικά και πολύ πιο αποτελεσματικά. Χρειάζεται λοιπόν να ε, δούμε πώς θα βοηθήσουμε τις περιφέρειες που είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση από αυτές που πραγματικά είναι οργανωμένες στο πεδίο της έρευνας και της τεχνολογίας. Χρειάζεται σίγουρα ε, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τη μείωση του προσωπικού. Πολλές περιφέρειες σήμερα δεν έχουν προσωπικό καν για να κάνουν το στοιχειώδη σχεδιασμό που χρειάζεται για την επόμενη προγραμματική περίοδο δεν υπάρχει το ανθρώπινο προσωπικό να οργανώσει διαβούλευση, να σκεφτεί με νέες ιδέες. Επομένως θα κάνει copy-paste, αντιγράψει κάποια άλλα σχέδια ή κάποιες παλιές ιδέες που ξεκίνησαν να συζητιόνται 10-20 χρόνια πιο πριν. Και αυτά που έχουν ξεμείνει από προηγούμενες περιόδους θα τα προτείνει να μπουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Δεν θα έχει καταλάβει ποιο είναι το, νέο πλαίσιο του κανονισμού για το Ταμείο συνοχή ή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή ανάπτυξη που πριν από λίγο ψηφίσαμε του κανονισμού. Ε, το λέω γιατί είμαι περιφερειακό σύμβουλο και βλέπω πώ σκέφτονται. Δηλαδή τα παλιά έργα που δεν είχαν ενταχθεί κάπου, αυτά τα έργα θα προτείνουν για την επόμενη περίοδο. Δηλαδή σκεφτείτε έργα που σχεδιάζονταν 10 χρόνια πριν, θα είναι αυτά που θα προταθούν για την επόμενη δεκαετία. Πώς θα προλάβουν να κάνουν καταγραφή των αναγκών να προτείνουν καινούριε ιδέε. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Μετά ένα δεύτερο πρόβλημα είναι το θεσμικό πρόβλημα. Πώ τα κράτη θα πιστούν ότι και η έρευνα πρέπει να αποκεντρωθεί. Αλλά ποιο φορέ μπορεί να κάνει έρευνα σήμερα είναι ένα ερώτημα. Τα ερευνητικά κέντρα είναι κυρίω τα πανεπιστήμια, είναι ειδικά ερευνητικά κέντρα. Ποιο μπορεί να κάνει έρευνα και ποιο μπορεί να μπει ακόμα και σε ευρωπαϊκέ χρηματοδοτήσει αν δεν είναι αναγνωρισμένο ω ερευνητικό κέντρο. Πόσες όμως περιφέρειες έχουν ερευνητικά κέντρα στην περιοχή τους. Συνήθως αυτά είναι σε, μεγάλες, σε πιο πλούσιες περιοχές ή σε μεγάλες πόλεις. Μικρές περιφέρειες ή αδύναμες περιφέρειες δεν έχουν ερευνητικά κέντρα. Επομένως ποιος θα ασχοληθεί. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Η οικολογική γεωργία στον νησιωτικό χώρο ή στον ορεινό χώρο. Ένα πανεπιστήμιο που κάνει αντίστοιχη έρευνα για τη γεωργία θα ασχοληθεί με τους μεγάλους κάμπους. Εκεί που υπάρχει πραγματικά το μεγάλο ποστό της αγροβιομηχανικής καλλιέργειας δεν θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα χαρακτηριστικά περιοχών. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε εκεί ακριβώ στον τομέα που λέμε τώρα εξειδίκευση ευφυή, σημαίνει ότι κάποιοι πρέπει να ασχοληθούν με ένα τομέα που αφορά μικρή περιοχή ή λίγου ανθρώπου. Και εκεί έχουμε, έχουμε βέβαια μια εμπειρία, οι κοινωνίε είχαν εμπειρίε, αλλά ήταν εμπειρίες, δεν ήταν επιστημονική έρευνα, αξιοποιούσαν την εμπειρία, τη σοφία, την παρατήρηση. Εμεί θέλουμε τώρα αυτά τα πράγματα συνδυαστούν και με επιστημονική έρευνα. Και υπάρχει πάντο κίνδυνο να έχουμε μία ανακύκλωση ιδεών και προτάσεων. Δηλαδή όσο πιο πολύ δυσκολεύει η εποχή, όσο πιο πολύ περιορίζει η πόρη, το ανθρώπινο δυναμικό, τόσο πιο πολύ είναι πιθανό να έχουμε ανακύκλωση παλιών ιδεών. Θα έλεγα ότι μαζί με τα πανεπιστήμια και με του επαγγελματικού και κοινωνικού φορεί πρέπει να δώσουμε έμφαση να αποτελέσουν ένα παράγοντα έρευνας και ένα παράγοντα που θα βοηθήσει σε αλλαγές ε, οι νέοι άνθρωποι που είναι σήμερα έχουν περάσει από σπουδέ, έχουν κάνει τα πτυχιακά, έχουν γνώσει, αλλά στην πραγματικότητα είναι άνεργοι. Δεν είναι δηλαδή καθιερωμένα ερευνητικά κέντρα, αλλά είναι νέοι οποίοι έχουν τη γνώση, αλλά είναι εκτό κοινωνική και επιστημονική εξέλιξη. Και εδώ πρέπει να δούμε ευέλικτα εργαλεία και από άλλε χρηματοδοτήσει, αλλά και μέσα από ερευνητικά προγράμματα, πώ μπορούμε κομμάτι αυτών των νέων που είναι σήμερα αν και είναι πάρα πολλοί, να μπορέσουν να δώσουν μια νέα όθηση στις ιδέες, στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και στην κοινωνική ανάπτυξη και καινοτομία. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Μην ξεχνάμε, ότι μόλις πριν λίγο συζητάγαμε για το e-health, αυτά τα πράγματα λοιπόν θα μπορούσαν να βασιστούν σε νέους ανθρώπους που έχουν πολύ καλή γνώση της πληροφορικής τεχνολογίας, ξέρουν δηλαδή, μπορεί να είναι γιατροί, αλλά μπορούν να εκπαιδευτούν και στη χρήση συστημάτων ε, ε, πληροφορικής τεχνολογίας. Πρέπει όμως να βρούμε κατάλληλα εργαλεία χρηματοδότηση που θα δώσουν νέα όθηση για να μπορέσουμε να μιλάμε μετά για ευφυή εξειδίκευση των περιφερειών, τουλάχιστον αυτών των περιφερειών που είναι σε μεγάλη απόκληση άσχετα από το ΑΕΠ του. Το ΑΕΠ δεν περιγράφει πάντα την πραγματική εικόνα, το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά πρέπει να δούμε τέτοια εργαλεία. Θα έλεγα καταλήγοντα μερικέ προτάσει. Ε, η επιτροπή μας θα πρότεινε να προσκαλέσει δύο περιφέρειες που έχουν μεγάλη εμπειρία και είναι πετυχημένα καλά παραδείγματα και δύο άλλες περιφέρειες που δεν έχουν καταλάβει καν ότι και το θέμα έρευνα και τεχνολογία αφορά και τις ίδιες. Δηλαδή να δούμε και από κοντά αυτή την απόκληση που υπάρχει και να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Ένα δεύτερο είναι ότι βέβαια δεν αφορά τόσο εμάς αλλά ίσως θα αφορούσε την, ε, ε, τον Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης μια συστηματική ενημέρωση των περιφερειών πάνω στα θέματα τη έρευνα. Συνήθω αυτό που κάνουν είναι να φτιάχνουν μια τέλειωτη λίστα με φορεί και να δημιουργούν ένα συμβούλιο καινοτομία, αλλά απλώ κάνουν ένα κατάλογο φορέων οι οποίοι θα καταθέσουν προτάσει. Όμω, σπάνια είναι ενημερωμένοι ακόμα και για τα υπάρχοντα εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή τι δυνατότητε συνεργασία. Άρα να προτείνουμε και στον Επίτροπο ε, μια τέτοια συνάντηση με εκπροσώπους των περιφερειών ώστε να αντιληφθούν ότι είναι διαφορετικό το πράγμα, διαφορετικά τα πράγματα σήμερα στο, θέμα της έρευνας και τεχνολογίας. Και φυσικά να, χρειάζεται να δούμε και συνέργειες με άλλες ε, επιτροπές όπως της απασχόλησης ε, και φυσικά και πολλές άλλες περιοχές και του περιβάλλοντος θα έλεγα ε, και βέβαια της Ήτρε για τα θέματα πώς μπορεί να υπάρχει μια συνοχή μεταξύ αυτών των πολιτικών. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία που έχει ε, που παρουσιάστηκε πριν. Φαντάζομαι ότι θα στήσουμε και άλλες ιδέες όταν θα ε, δουλέψουμε πάνω σε αυτή πιο αισθηματικά. Αλλά νομίζω ότι ε, είναι αυτό, να σκεφτούμε καινοτόμε ιδέες και εμείς ως ευρωπαϊκός θεσμός για να βοηθήσουμε τις φορείς που έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Γιατί αυτό που πολλές φορές διαπιστώνει κανείς είναι ότι προχωρούν ορισμένες περιφέρειες, ορισμένοι φορείς μπροστά και καλά κάνουν, αλλά πίσω μεγαλώνει η απόσταση, ειδικά τώρα την περίοδο της κρίσης και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Ευχαριστούμε, Νίκο. Υπάρχει κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτια Ρέπελ, καλώς ήρθατε. Τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να σας ευχαριστήσω που φύγετε το θέμα αυτό της στρατογικών ευθύους εξειδίκευσης με μια συγκεκριμένη έκθεση εφηρεωμένη στο θέμα. Μετά τη μεγάλη στηρίξη που είχαμε από το Ευρωκοινοβούλιο για την πρόταση κανονισμών για την εξάντερη και επειδή αυτό συζητήθηκε και κατά τους τριμμένους διαλόγους και τις διαπραγματεύσεις, έζησε το μικρόφωνο μου, τώρα αυτό λαμβάνει τη μορφή έκθεσης. Τέθηκε ερώτημα για το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης, προσωπικός. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να είχαμε ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα, αλλά σε καμία περίπτωση ποτέ δεν είναι αργά. Στο τέλος αυτής της χρονιάς ή στην αρχή της επόμενης, τα λειτουργικά προγράμματα των ευθυνών στρατηγικών εξειδικευσής δεν βρίσκονται στο τέλος τους, αλλά στην αρχή τους. Θα είναι το ξεκίνημα. Ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα είναι μία προσπάθεια συμπλήρωσης ε, κοιτίων για να μπαίνει ένα τσεκ, αλλά ότι θα ξεκινήσει η φάση υλοποίησης των στρατηγικών στην πράξη, στην πραγματικότητα θα ξεκινήσουν, δηλαδή θα ξεκινήσει αναζήτηση σχέσεων συνεργασίας με άλλες περιφερειές και άλλα κράτη προκειμένου να υπάρξει βελτίωση και περισσότερες ακριβώς ε, συνδυαστικέ προσπάθειες λόγω και του περιορισμού δημοσίων κονδυλίων πανευρωπαϊκά. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε ωφέλη από την ε, συνεργασία και την αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει να τονώσουμε το δυναμικό ε, κοινών προσπαθειών ε, ανά την Ευρώπη. Και μια μικρή επικριτική παρατήρηση. Κάποιες φορές δεν επικεντρώνονται οι περιφέρειες στο τι συμβαίνει αλλού. Επικεντρώνονται πολύ στο δικό τους χώρο και στο τι γίνεται από οικονομικής άποψης, με τα κονδύλια. Πρέπει να ανοίξουν λίγο τα μυαλά και των περιφερειών ε, και να ανοίξουν οι ορίζοντές τους. Αυτό είναι κάτι που το καλωσορίζουμε ως ε, πρόταση. Και μια-δυο παρατηρήσεις. Δεν έχω απαντήσεις σε όλες τις ιδιαίτερα εύστοχες ερωτήσεις που έχουν πεθεί στην έκθεση, αλλά ήθελα σε κάποιες να σταθώ. Ο τελευταίος ομιλητής πολύ ορθός, ρώτησε εάν αφορά αυτό όλες τις περιφέρειες ή ενδεχομένως ένα μικρό όμιλο, ένα κλαμπ των καλύτερων, μια ελίτ με, που διαθέτουν ήδη τα μέσα για την ε, καινοτομία. Πίσω από τη στρατηγική ευθύου εξειδίκευση ε, και την έννοια αυτή υπάρχει ακριβώ η σκέψη να ανοίξουμε την πόρτα σε περιφέρειες που ω τώρα δεν υπήρξαν αρκετά καινοτόμε. Δεν έχουν αξιοποιήσει το δυναμικό καινοτομία που διαθέτουν στο μέγιστο βαθμό. Όπω είπατε, δεν αφορά μόνο την τεχνολογική καινοτομία η προσπάθεια αυτή, αλλά πρέπει να σκεφτούμε εφάντα τους τρόπους για να ξεκινήσουμε προσπάθειες προσπάθειες πραγματικής ανανέωσης των δράσεών μας και να προκύψουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εστιάζουμε λοιπόν και σε περιφέρειες που δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά και πιστεύουμε ότι μπορούν να προκύψουν καινοτόμε ιδέες και η κατάλληλη χρηματοδότηση για αυτές. Επίσης τέθηκε ένα ερώτημα για την διάθεση των ε, δεδομένων, των στοιχείων και το πόσο υπάρχει δυσκολία να συνδυαστεί το Horizon 2020 με τα διευθυντικά ταμεία. Η δυσκολία είναι να εκπονηθούν στρατηγικές που να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτές τις προτεραιότητες. Προφανώς αυτό δεν είναι ένα απλό εγχείρημα. Το γνωρίζουμε καλά και σημειώσαμε ότι από τις περιοχές 200 συν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στις πλατφόρμες για τη συγκέντρωση στοιχείων αυτής της Εβίλης που θέλει να εξυπηρετήσει τα κάτι μέλη και τις περιφέρειες. Ε, είναι αλήθεια αυτό, αλλά ήταν ε, εθελοντική η διαδικασία. Δεν πιέσαμε τα κάτι μέλη να συμμετάσχουν, αλλά με ενδιαφέρον είδαμε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία περιφερειών πάρα πολλέ περιφέρειε, διαφορετικέ μεταξύ του, που θέλουν να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική αρχή. Τα καλά νέα είναι ότι ω τώρα 140 περίπου περιφέρειες από τα κράτη-μέλη συμμετέχουν σε αυτή την πλατφόρμα και 9 κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο ε, έχουν προσχωρήσει επισήμω. Δεν ήταν απλό το εγχείρημα, όπω είπα. Αλλά παίρνοντα αφορμή από τι παρατηρήσει για τα νησιά, τα ορεινά μέρη, τι απομακρυσμένε περιοχέ, τι απομονωμένε περιοχέ, πέραν της πλατφόρμας αυτής που είναι ανοιχτή για όλους και συνδυάζει τις προσπάθειες διαφορετικών περιφερειών, δίνεται ίσως και η ευκαιρία σε παρόμοιες περιοχές να συζητήσουν παρόμοια προβλήματα και να δουν στην πράξη τι συμβαίνει ή να σκεφτούν από κοινού πρακτικές λύσεις. Συχνά προσφέρουμε και τη δυνατότητα να γίνονται εξ, εξαγωγές Ω τώρα είχαμε τουλάχιστον 90, ε, μάλλον, 90 ε, συμβάσει είχαμε τώρα για την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων σε, 70 περιφέρειες από 19 κράτη-μέλη. Έτσι τονώνεται η εξειδίκευση και καλλιεργείται η εξειδίκευση στις περιφέρειες συγκεκριμένα. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι συμφωνώ απολύτως ότι υπάρχει ανάγκη να συμμετάσχουν εδώ διαφορετικές γενικές διευθύνσεις, ίσως και διαφορετικές ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας και των ε, μεταφορών. Είναι μια ε, διαδικασία διατομιακή. Θα μπορούσε λοιπόν η περιβαλλοντική πολιτική να συνδυαστεί με την βιομηχανική και όλοι οι πολιτικοί ηθήνοντες να συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για αυτή την πρόταση. Πρόεδρος και εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση για την πλατφόρμα. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να το λόγο. Ο Λαμπέρτ. Ευχαριστώ. Θα συναντηθούμε με εθνικούς βουλευτές. Το Νοέμβριο είναι. Ναι, το Νοέμβριο. Δεν θα ήταν μια ωραία έκπληξη να τους ενημερώσουμε για αυτά και ο κύριος Βίνκλερ ίσως μπορεί να βοηθήσει. Γιατί, γιατί εγώ είχα μια συνάντηση με τον κύριο Μαρινέσκου, τον Ρουμάνο συνάδελφο από την ομάδα μας και με κάποιους εκπροσώπους περιφερειών από την Ρουμανία. Και ήταν σε μια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Μα τι λέτε, μα είπανε. Δεν έχουμε ιδέα. Κανείς δεν έχει ζητήσει τη γνώμη μας. Οπότε δεν μπορείτε να κατηγορήσετε τις περιφέρειες που δεν είναι ενημερωμένες ή ακόμα τους εθνικούς βουλευτές που δεν έχουν ιδέα για το περίφημο S3, τις στρατηγικές δηλαδή ευθύους εξειδίκευσης. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα. Ναι, Λαμπέρ, συμφωνήσαμε να αναφερθούμε στις προκλήσεις της επόμενης περίοδου. Οπότε, ναι, μπορεί κάλλιστα να συμπεριληφθεί. Ευχαριστώ να το συμπεριλάβουμε. Και πριν ε, σας δώσω το λόγο πάλι, Χέρμαν, μίλησα με τον Βικέλ και μπορούμε να επιταχύνουμε κάπως την όλη διαδικασία από ό,τι φαίνεται, γιατί η έκθεσή σας έχει προχωρήσει. Θα δείτε, μιλήστε με τη γραμματεία για να δούμε αν θα διατηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα ή θα επιταχύνουμε. Θέλετε και εσείς το λόγο τώρα, παρακαλώ, για να κλείσουμε. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, για όσα μου είπαν και αυτά που είπε και η Κομισιόν. Υπάρχουν φυσικά ακόμη πολλά θέματα που είναι ανοιχτά και μπορούμε να τα απαντήσουμε μόνο από κοινού γιατί οι ερωτήσεις ε, δεν υπάρχουν ακόμη, δεν τις έχουμε. Και οι συνάδελφοι ε, είπαν σαφώς ότι χρειάζονται συμβουλές. Δεν ε, είναι βεβαίως πανάκι αυτό για όλα. Βεβαίως πρέπει να δώσουμε αυτή τη βοήθεια και για το δεύτερο. Νομίζω ότι και εσύ το έθεσες πολύ σωστά, Λάμπερτ. Μας φτάνει ο χρόνος. Μήπως πρέπει να διαπραγματευτούμε με τα κράτη-μέλη. Βεβαίως είναι λίγο περιορισμένος ο χρόνος. Αλλά θα τα καταφέρουμε αν καταλάβουν οι ε, περιφέρειες ότι πρέπει να προωθήσουν και να εξελίξουν περαιτέρω την στρατηγική τους. Και ίσως θα πρέπει να έχουμε και ένα σύστημα επιτήρησης για να υπάρξει η περαιτέρω καταγραφή της στρατηγικής τους συγκεκριμενοποίησης και αν το καταφέρουμε από κοινού, τότε είμαι αισιόδοξο ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να πάρουμε αποφάσει σήμερα. Απλώ για να έγγραφο εργασία πρόκειται. Την επόμενη φορά θα ακούσουμε και το σχέδιο έκθεση και θα δούμε αν θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε ή όχι. Ωραία. Έτσι λίγη και αυτό το θέμα. Σα ευχαριστώ όλους. Οι συντονιστέ τώρα παρακαλώ, γιατί έχουμε αμέσω τώρα τη συνεδρίαση των συντονιστών. Έχουν εξαφανιστεί κάποιοι, μήπως οι βοηθοί μπορούν να τους βρούνε. Αλλιώ να φωνάξω την αστυνομία, αλλά. Να, ήδη έχουμε εδώ την κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ. Κατά τα άλλα, αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε στις 9.